Thank you, friends. Καλησπέρα σας. Κάποιοι χρειάστηκε να τρέξουν για να φτάσουν στην ώρα τους. Λοιπόν, καλώς ήλθατε. Η κυρία Βεραγιουροβά, αντιπρόεδρος για αξίες και διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάντοτε καλοδεχούμενη. Μας τιμά η παρουσία της και στο πάνελ για τον λεγόμενο διαστρωμένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το πρώτο θέμα μας, το οποίο αφορεί την ε, ελευθερία των μέσων της αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κρατός δικαίου, στην περιλαμβανομένη της ετήσιας έκθεσης προηγή της, του χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και, και εξαρτήσει του κατά πόσον θα προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, Σύμβαση για τα του Ανθρώπου. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 6 της ε, συνθήκης, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη. Ε, άλλες ευθύνες που έχει η κυρία Γιουρόβα και τα οποία θα συζητήσουμε, άλλο με το ενδιαφέρον, και τα χέρια που θα δω να σηκώνονται. Αλλά ας δώσουμε τον λόγο πρώτα απ' όλα στην Αντιπρόεδρο και μετά θα περάσουμε σε συζήτηση ξεκινώντα με τους συντονιστές και μετά με τους υπολείπους. Όμως, όπως το λέω συνεχώς, μην ξεχνάτε ότι είναι από τις φορές που πραγματικά πιεζόμαστε από χρόνο. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο πάνελ. Είχαμε έξι ομιλητέ και μετά συζήτηση. Από μια μισή ώρα ο καθένα προφανώ δεν μα έφτασε. Το ίδιο και απόψε. Μια μισή ώρα πάντω είναι το όριο για, την, για τον πρώτο γύρο τη συζήτηση με την κυρία Γιώργα. Σίγουρα δεν είναι αρκετό, αλλά όταν δείτε ότι πλησιάζουμε στο όριό μα, να θυμάστε ότι έχουμε και έναν δεύτερο αντιπρόεδρο, τον κύριο Σχοινά, για την ε, πρόθεση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωή. Λοιπόν, ξεκινούμε, κυρία Γιώργα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο χρόνο είναι σημαντικό, το ίδιο όμω και η διαφάνεια και οι αξίε. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, που επανέρχομαι δηλαδή. Η πρώτη ευκαιρία να μιλήσουμε. Είναι και μια σημαντική ευκαιρία να ξεκινήσει η νέα μας θητεία. Όπως γνωρίζετε, με πολλούς από εσά έχουμε συνεργαστεί στην προηγούμενη θητεία. Ευχαριστώ γι' αυτό. Σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν επί των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με την ίδια ζέση. Η ζήτησή μας λαμβάνει χώρα σε στιγμή γιατί μόλι η Κομισιόν δημοσίευσε ψηφιακό πακέτο Ακριβώ για την αντιμετώπιση μια πολύ σημαντική απειλή, προ, ε, πρόκληση μάλλον τη εποχή μα την ψηφιακή επανάσταση. Συζητούμε θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα προσφυλή στην Επιτροπή, η αξιόπιστη μεταξύ άλλων μεταφορά δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Με βάση αυτό το πακέτο, αυτή τη δέσμη, θα μιλήσουμε και για το τρίπτυχο που μας είναι ιδιαίτερως προσφυλές, δηλαδή κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα και δημοκρατία. Η ψηφιακή αυτή δέσμη που εγκρίνουμε και συζητούμε σήμερα κρατείνει στο ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι αντιστρόφως. Και αυτό είναι μια ένδειξη αυτού που θέλουμε να πετύχουμε ως ευρωπαϊκό μοντέλο βάσει της αριστείας και της εμπιστοσύνη. Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο είναι απολύτως συμβατό με τις αξίες μας και τις αρχές μας και το οποίο εδράζεται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο είναι κατά των διακρίσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό από την αρχή. Η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει, αναδιαμορφώνει τα πάντα την οικονομία μεταξύ άλλων, όμως γύρει και ζητήματα που αφορούν την ανθρωπίνη αξιοπρέπεια, την ιδιωτικότητα, την καταπολέμηση των διακρίσεων, τη διαφάνεια κλπ. Στη λευκή βίβλο που δημοσιεύσαμε σήμερα αναλύεται η πολιτική περί των κανονιστικών και άλλων εργαλείων για να επιτευχθούν οι δύο στόχοι. Πρώτον, η προογή της, η προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποίηση με σεβασμό αυτών των νέων τεχνολογιών. Η διαβούλευση θα συμβάλλει στην, ε, στις μελλοντικές αποφάσεις της Κομισιόν. Αξιολογούμε τον κίνδυνο για παιδεία υψηλού κινδύνου, υγεία, αστυνομία, μεταφορές, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί θέλουμε ίχνη λασιμότητα και τον τελικό λόγο να τον έχουν οι άνθρωποι. Για τις σχετικές εφαρμογές Επίσης η Κομισιόν προτείνει ένα σύστημα σήμανσης. Δεν θέλουμε τα λεγόμενα μαύρα κούτια, τα οποία δεν μπορούν να τύχουν πλήρους επιβλέψης. Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης επί των κοινών μας αξιών μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάποια στιγμή, όμως η αξιοπιστία, όπως είπα, είναι πολύ σημαντική για την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών και της χρήσης τους. Η σημερινή ψηφιακή δέσμη περιλαμβάνει και πολιτική για τα δεδομένα. Η ισχύ μα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή δράζεται στην εσωτερική αγορά και αυτό πρέπει να φροντίσουμε και για τα δεδομένα. Χρειαζόμαστε καλύτερους τρόπους ανταλλαγή και αξιοποίηση δεδομένων και δι των βιομηχανικών. Προ το σκοπό αυτό να μην ξεχνούμε την παγκόσμια διάσταση. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ιαπωνία και άλλους εταίρους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο για να προαγάγουμε την ανταλλαγή δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις. Εάν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, θα καταλήξουμε, πιστεύω, στην κατάλληλη νομοθεσία και θα είμαστε πρωτοπόροι πλέον στην ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως κάναμε και σε άλλους τομείς στο παρελθόν. Ας δούμε τώρα τα άλλα βασικά θέματα της εντολής μου κράτος δικαίου. Θα είμαι σαφής. Το κράτος δικαίου είναι θεμέλιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι γίνεται σεβαστό παντού και πάντα και ότι όλες οι χώρες την χάνουν ισότιμης μεταχείρισης. Η Κομισιόν έχει αναλάβει σχετική δράση στο παρελθόν και θα το ξανακάνει αν χρειαστεί βάσει των κοινών αξιών και βάσει της νομοθεσίας. Ας μην ξεχνούμε ότι η τήρηση του κράτου δικαίου δεν είναι μόνο καθήκον της Κομισιόν. Είναι κοινή υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, των κρατών μελών και βεβαίω της Κομισιόν. Το έργο μα. εν είναι διτό. Θέλω να επιβεβαιώσω σήμερα ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των συνθήκων, εάν η νόμοι που ψηφίζονται σε μια χώρα δεν είναι συμβατοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να δρομολογήσουμε τι σχετικέ διαδικασίε όπω προβλέπεται από την σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αξιοποιώντα όλα τα εργαλεία, σαρτήσει συμπεριλαμβανομένε τι διαδικασίε παραβάση. Συζήτησαμε το θέμα στην προηγούμενη Ολομέλεια. Αξιολογούμε αυτή τη στιγμή την πειθαρχική νομοθεσία στην Πολωνία. Έχουμε διατυπώσει τις σχετικές μας ανησυχίες και να είστε σίγουροι ότι δεν θα μασίσουμε τα λόγια μας εάν καταλήξουμε στο σχετικό συμπέρασμα. Δεύτερον, η Κομισιόν εργάζεται για ένα νέο εργαλείο πρόληψης που αφορά την δημιουργία, την θέσπιση ενός ετήσιου κύκλου παρακολουθήσεις των θεμάτων κρατούς δικαίου στις χώρες μας για να επιβεβαιώνουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη δυνατότητα αντιμετώπισης της διαφθοράς και της προστασίας των μέσων. Θα μελετήσουμε τις μεθόδους συλλογής δεδομένων στα κράτη-μέλη. Σκοπός μας είναι να δημοσιεύσουμε τα σχετικά στοιχεία το φθινόπωρο μετά από συζήτηση με εσάς και με το Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή, η αίτηση αυτή αναφορά, πιστεύω ότι θα βελτιώσει τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τα θέματα κρατού δικαίου, είμαι στη διάθεσή σα για να συζητήσουμε οτιδήποτε σα ενδιαφέρει. Αυτό ήταν και ο βασικό λόγο της επισκεψή μου στην Βαρσοβία. Γιατί σκοπό μα είναι να παραμείνουμε κοινότητα αξιών και αρχών, αλλά και κοινότητα διαλόγου. Τέλος, καθώ πλησιάζει το ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τον Ευρωπαίο φορολογούμενο στα πλαίσια ε, του κράτους δικαίου. Χαίρομαι ότι το θέμα παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να ξέρετε ότι θα καταψηφίσω οτιδήποτε αποτελεί ταπείνωση του επίπεδου των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δέκα χρόνια μετά από την έγκριση του σχετικού χάρτη θα συνεχίσω να προσπαθώ για την αναθεώρηση αυτής της πολιτικής. Θέλω να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στα θέματα εφαρμογής ή επιθεμάτων όπως η απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και για την εφαρμογή του χάρτη σε επίπεδο κράτους μέλους. Στο πλαίσιο αυτό είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ξεκινούμε και πάλι τις διαβουλεύσεις για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όπω γράφω στην σχετική επιστολή μου, θα έχω τη χαρά να σας ενημερώνω τακτικότητα, ώστε να παρακολουθείτε και εσείς σε πολιτικό επίπεδο διαβουλεύσεις. Και ο τρίτο πυλώνας, η δημοκρατία. Εδώ θέλω να καταθέσω ορισμένε σκέψει σχετικά με το σχετικό σχέδιο δράσης. Πρόκειται για απόκριση σε πολλές προκλήσεις για τη δημοκρατία μας, όπως οι περισφυρσίε σε διαδικασίες εκλογικές ή οι παρεμβάσει στην ελευθερία των μέσων. Ξέρετε, δεν κινούμε επί μηδενική βάσεως. Υπάρχει ένα μια δέσμη μέτρων για τις ε, εκλογές. Ε, θα τα αξιολογήσουμε όλα αυτά και θα προχωρήσουμε. Ίσως ε, μάλιστα να εξετάσουμε και το δεχόμενο λήψης νομοθετικών μέτρων ή κανονιστικών μέτρων. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε τους μέσο κατά πλατφορμών που με βάση συγκεκριμένους αλγορίθμους επηρεάζουν την ελευθερία των μέσων και θα εργαστούμε και θα εξετάσουμε τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων. Ξέρουμε επίση για τι απόπειρε χειραγώγηση των μέσων στο διαδίκτυο με χακάρισμα ε, τύπου Cambridge Analytica. Θέλουμε λοιπόν να παρακολουθούνται τα μέσα αυτά και από τα κράτη-μέλη. Ε, είδα τη Δευτέρα τον Σούκεμπερ και του είπα ότι Ξέρουμε ότι οι πλατφόρμες μέσω κοινωνική δικτύωσης βοήθησαν. Τώρα θέλουμε να υπάρχει στον τομέα αυτών περισσότερη ευθύνη και περισσότερη λογοδοσία. Η δέσμη, μάλλον το σχέδιο δράση αφορά και τα μέσα. Στην προσεχή σύνοδο στις 15 Μαρτίου θα συζητήσουμε τα ευρήματα της έρευνας για τον πλουραλισμό των μέσων. Είμαι σίγουρος ότι τα στοιχεία αυτά θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όμω, για να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση χρειαζόμαστε περισσότερα. Το ψέμα είναι σοβαρό. Το πιο σοβαρό είναι όμω ότι ο κόσμος πιστεύει αυτά ψέματα. Η συνεργασία λοιπόν με τα κρατημέλη και τις πλατφόρμες πρέπει να καταλήξει περισσότερη δύναμη στα χέρια των πολιτών. Να ενημερώσουμε περισσότερο του πολίτε σχετικά με τα μέσα, για το πώ λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες, να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση και παράλληλα να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας να εντοπίζουμε το ταχύτερο δυνατόν τις ψευδοειδήσεις. Θα μιλήσω με την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης, την Stratcom και το ΝΑΤΟ για το θέμα αυτό. Θα συζητήσω τα ζητήματα αυτά επίσης κατά τη διάρκεια της προσεχού επισκεψή μου στι ΗΠΑ, δεδομένου ότι και εκεί έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το πώ αντιμετωπίζει κανεί την παραπληροφόρηση. Ε, Κατακλείδη και συμπερασματικά θα ήθελα να καταθέσω την ετοιμότητά μου και την πρόθεσή μου να συνεχίσω να συντονίζω τα θέματα δικαιοσύνη, διαφάνεια, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα, την προστασία των δεδομένων τα οποία πολλούνται ει βάρο των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να καλέσω του βουλευτέ αυτή τη επιτροπή να καταθέσουν τι δικέ του απόψει επίση για την εξέλιξη του φακελού GDPR για την περαιτέρω εφαρμογή με παραλή υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επίση κάτι πολύ σημαντικό με έναν τρόπο συνεκτικό παρά με τροποποίηση τη σχετική νομοθεσία. Περιμένω τι ερωτήσει και τα σχόλιά σα και προσβλέπω σε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή σας καθώς και με την ε, προσωρινή Επιτροπή για την παραπληροφόρηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θέσατε επιτάπητος πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και η Επιτροπή Πολιτικών ε, Ελευθεριών ασχολείται με τη δημοκρατία το, και το κράτος δικαίου. Η Υπάρχουν πολλά εκρεμή ζητήματα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας αρχίσουμε τη συζήτηση πρώτα με τους συντονιστές. Ο κύριος Λένερς έχει το λόγο. Δύο λεπτά για τον κάθε συντονιστή, έτσι ώστε να μπορέσετε να λάβετε το λόγο όλοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισήγηση σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και το ψηφιακό μέλλον. Έχει μεγάλη σημασία το τεχνολογικό μέλλον των ανθρώπων και η ενιαία αγορά. Αυτό αφορά και τις δημοκρατικές αξίες. Έχουμε τη Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη και υπάρχει και ένα ε, σχέδιο, ένα πρόγραμμα για το, τρίτο, για το τέταρτο τρίμηνο. Νομίζετε ότι έχουμε επαρκή, επαρκές χρονικό διάστημα ή χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο χρόνο. Ως προς το πρόγραμμα δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, διότι είμαστε πέραν της ιδέας ε, της ε, θελούσιας συμμετοχής, ιδιαίτερα ως προς τις τεχνολογικές πλατφόρμες. Αν θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία, τότε θα πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο ως προς τη διαφάνεια των αλγορίθμων, τουλάχιστον για την πρώτη φάση του εγχειρήματος. Ε, είχαμε και τον γενικό, την Γενική Εισαγγελέα, την Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελέα εδώ, που μας μίλησε για το ότι δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε την απάτη αν έχουμε εισαγγελείς με μερική απασχόληση μόνο. Ε, οι αξιωματούχοι δεν είχαν κάτι να προσθέσουν. Ίσως μπορείτε να μας απαντήσετε εσείς, διότι το ζήτημα το σημεριζόμαστε. Και εδώ, σε σχέση με την ετήσια έκθεση του κράτους δικαίου στο δεύτερο εξάμεινο, πώς προβλέπετε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς τα θεσμικά όργανα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν δυνάμει της διαδικασίας του άρθρου 7. Βλέπετε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκτός μικροφώνου ο Προεδρεύων, κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε την Επίτροπο Γιούροβα που τουλάχιστον αναφέρθηκε σε όλα τα σημεία. Υπάρχει ένα πολύ ευρύ χαρτοφυλάκιο εδώ. Θα ήθελα να σταθώ στους τρεις πυλώνες κράτος δικαίου, δημοκρατία και θεμελιώδη δικαιώματα και οι τρεις ε, πυλώνες θα πρέπει να συνυπάρχουν. Αλλά υποβάλλω το ερώτημα γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η κοινή γραμμή Επιτροπής Κοινοβουλίου. Αλλά δυστυχώς το πρόβλημα έγκυται στα κράτη-μέλη, στο Συμβούλιο. Ακόμα και στο επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων η Ουγγαρία και η ε, Πολωνία δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Άρα τι νόημα έχει να προωθούμε νομοθεσία, συγκεκριμένη νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τον συνδυασμό του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την τήρηση των αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εάν τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει, θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτά τα πλαίσια. Νομίζετε ότι μπορείτε να πιέσετε περισσότερο τα κράτη-μέλη για βελτίωση της κατάστασης θα ήθελα να επανέλθω στην τεχνητή νοημοσύνη και την συνεργασία, τον επιμερισμό και την συμμετοχή στα δεδομένα. Όταν πρόκειται όμως για κοινή συμμετοχή στα δεδομένα, όταν συνδυάζουμε τις διάφορες πηγές, ίσως το τέλος φτάνουμε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Άρα δεν τίθεται θέμα τεχνητής νοημοσύνης μόνο, αλλά το πώς χτίζουμε νέες ιδέες πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και την ε, προστασία των δεδομένων έτσι ώστε να έχουμε ανώνυμα στοιχεία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την διαφάνεια. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων και με τον Επίτροπο Βέστερ γιατί θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και να ταυτοποιούμε τα στοιχεία που πραγματικά μας βοηθούν. Δεν είχα χρόνο να διαβάσω το έγγραφο που εκδόθηκε σήμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ μαζί μας. Ιντβέλτ, ευχαριστώ, ε, χαίρομαι που είστε εδώ Επίτροπε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπατε και η πολιτική ομάδα Renew θα σας στηρίξει έτσι ώστε να δράσουμε τάχιστα. Μπορεί να υποθεί το ίδιο για την κυρία Φαντελάιεν ε, θα σας υποστηρίξει όταν θα πρέπει να λάβετε μέτρα κατά της Ουγγαρίας ή της ε, Πολωνίας, γιατί είχε πει για την Πολωνία «Α, κανείς δεν είναι τέλειος». Αλλά αν δούμε πώς αποδομείται το κράτος δικαίου στην Πολωνία, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, γιατί κάθε μέρα που περνάει δημιουργεί ανήκε στο βλάβη και νομίζω ότι δρούμε χωρίς ευθύνη. Αυτό το βλέπουμε και στη Γερουσία με τους Ρεπουμπλικανούς. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα στεγανό μέτωπο για να υποστηρίξουν κάποιον που παραβιάζει το νόμο. Αυτό το βλέπουμε και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βλέπουμε ότι η αιρεσιμότητα έχει ήδη αποδυναμωθεί. Ως προς το πρόγραμμα δράσης υπέρ της δημοκρατίας θα ήθελα να δούμε τι κάνουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί που διαδίδουν ψευδείς ειδήσει, όπως τις επωνομάζουμε. Για παράδειγμα, ο κύριος Όρμπαν με τον αντισημιτικό του λόγο, με την ομοφοβία που προωθεί, έχει ένα κύρος. Μπορούμε να ε, καταγγείλουμε το Facebook, αλλά αν δεν μπορούμε να καταγγείλουμε πολιτικά κόμματα και πολιτικούς, τότε υποσκάπτουμε την δική μας ε, αξιοπιστία. Ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, συμφωνώ, καμία διάκριση να μην υπάρχει και να προστατεύονται τα δικαιώματα των προσώπων. Όταν όμως μιλάμε για προστασία των πολιτών, βρισκόμαστε πίσω έτη φωτός και με εκπλήσι που η Επιτροπή θα αποσύρει προτάσεις που στην ουσία προστατεύουν τους πολίτες ως προς την ιδιωτικότητά τους, τον κανονισμό περί διαφάνειας και ούτω καθεξής. Θα πρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει αυτές τις προτάσεις, γιατί έτσι οι πολίτες θα έχουν την προστασία που χρειάζονται. Ευχαριστούμε πολύ. Η πράσινη, η κυρία Στρίκ, η κυρία Ράνκε. Έχετε το λόγο. Ε, ζητώ συγγνώμη, θα μιλήσω στα γερμανικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Επίτροπε που είσαστε εδώ. Μιλάμε για την κατάσταση στην Πολωνία και μιλάμε και για διαφάνεια δυνάμει του άρθρου 7 καθώς και τη διαδικασία επί παραβάση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα ήθελα ορισμένες διασαφηνίσεις για την εκστρατεία μίσους από πλευράς Πολωνίας κατά συγκεκριμένων πολιτικών. Μιλήσατε και για το πολιετές, για το κράτος δικαίου και την αιρεσιμότητα. Νομίζω ότι θα Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι όταν μιλάμε για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια του προγράμματος των δικαιωμάτων και αξιών, θα πρέπει να εξασφαλίσετε την εφαρμογή αυτού του πλαισίου. Κάτι άλλο στο οποίο δεν αναφερθήκατε, τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε δραματικές εξελίξεις σε σχέση με την άκρα δεξιά και τη δράση της, τρομοκρατική της δράση στη Γερμανία. Ε, έγιναν, μάλλον υπάρχουν 402 εντάλματα συλλήψεων κατά μελών της άκρας δεξιάς και δυνάμει τρομοκρατών. Νομίζω ότι είμαστε παρατηρητές μόνο στη δράση αυτών των πυρήνων. Έχουμε δίκτυα τρομοκρατίας, τα οποία δεν αντιμετωπίζουμε. Βλέπουμε ότι ε, γίνονται επιθέσεις κατά τζαμιών, σαν να ζούμε μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και η Επιτροπή θα πρέπει να δει τι μπορεί να κάνει για να καταπολεμήσει αυτή τη μάστιγα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και θα ήθελα κάτι να κάνει η Επιτροπή. Ο κύριος Καρντίνο από το ID. Ο κύριος Φέστα, ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την κυρία Ράιντκε γιατί μίλησε για την τρομοκρατία στη Γερμανία. Ξέρετε πως τις τελευταίες ε, μέρες και πιο συγκεκριμένα προχθές η Ευρωπόλ ε, μίλησε για την τρομοκρατία που προέρχεται από τα αριστερά ως κύρια πηγή τρομοκρατίας εποχής μας. Ήταν στην Frankfurt είναι την εφημερίδα αυτή, για τις διασυνδέσεις μεταξύ αριστερής τρομοκρατίας, των αριστερών και των πράσινων. Οπότε, το κόμμα του κ. Κάρν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλές επιθέσεις από την αριστερά. Κυρία Γιούροβα, μπορείτε να ασχοληθείτε με το θέμα. Ξέρουμε πως στη Θουρυγγία οι φιλελεύθεροι δεν ε, θα είναι πλέον στην κυβέρνηση, αλλά τουλάχιστον να μην υποστούν υποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ για την ECR. Ε, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιάκη. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πολωνικά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο καταρχήν για τις δηλώσεις που έκανε για τη μελλοντική συνεργασία για το ποινικό δίκαιο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η Πολωνία έχει μειωμένα επίπεδα εγκληματικότητα ε, τα τελευταία χρόνια. Πέφτει η εγκληματικότητα ε, με πολύ ταχύ τρόπο, με τον ταχύτερο στην Ευρώπη και για το κράτος δικαίου να σου πω ότι είμαι 7 μήνες εδώ και μου λένε συνέχεια και ακούω συνέχεια πως δεν πάνε καλά τα πράγματα με το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Αλλά κανείς δεν μου λέει συγκεκριμένα τι δεν πάει καλά, ποιοι είναι οι νόμοι οι οποίοι στην Πολωνία ε, καταπατούν ε, τους ε, νόμους τους σχετικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι δηλαδή οι πολιτικοί διορίζουν τους δικαστές. Μα στην Πολωνία οι δικαστές επιλέγουν τους δικαστές. Αντίθετα, σε άλλα κράτη-μέλη είναι η πολιτική ηγεσία που διορίζει τους δικαστές τώρα. Ε, το πειθαρχικό δίκαιο του δικαστικού σώματος. Ποια ακριβώς παράγραφος ή διάταξη είναι αυτή που έρχεται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Να σας δώσω το εξή παράδειγμα. Στη Γερμανία, γιατί οι ίδιες παραβάσεις του δικαστικού μπορούν να κινηθούν και ποινικέ διαδικασίες κατά των δικαστών, ενώ αυτό τουλάχιστον στην Πολωνία δεν γίνεται. Άρα λοιπόν θεωρείται ότι αν κανείς διώκεται σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα υποφέρει πιο πολύ παρά αν διώκεται ποινικά. Μα αυτό αποκλείεται. Επίσης, το χειρότερο είναι το εξής. Σπέρνεις ψευδείς πληροφορίες. Συγγνώμη, το κάνετε εσείς για την Πολωνία. Αυτό γιατί πρέπει να γίνει δεκτό. Η κυρία Έρνστ. Είστε εδώ για να μας μιλήσετε για τις αξίες και για τη διαφάνεια. Αυτός είναι ο τίτλος του χαρτοφυλακίου σας. Να μας πείτε λοιπόν δύο λόγια για τη διαφάνεια, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό και είναι και σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή να έχουν την εντύπωση πως εμείς εδώ κάτι κάνουμε. Πως τα ενδιαφέροντά τους στηρίζονται. Επίσης, για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων και τους κανόνες σχετικά. Τι θα συμβεί με τα δεδομένα που αφορούν τους πολίτες μας όταν θα χρησιμοποιούμε περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Πώς θα σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα για το τι θα συμβεί και ακόμα πιο συγκεκριμένο όταν μιλάμε για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πώς μπορούμε αυτό να το ταιριάξουμε με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και το μέλλον προς το οποίο κινούμαστε. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια κομμάτια. Και μετά περνάμε και στην τρομοκρατία από την άκρα δεξιά. Ευρωπόλ μίλησε για κενά. Κενά στη δίωξη των τρομοκρατών από την άκρα δεξιά. Από το 1990 και μετά είχαμε 198 θύματα στη Γερμανία. Βεβαίως μπορούμε να το δούμε ε, από οποιαδήποτε σκοπιά και να χρηματοδοτήσουμε οποιοδήποτε πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι πέραν της τρομοκρατίας θα πρέπει να δούμε και το θέμα της άκρας δεξιάς. Και γι' αυτό ε, πρέπει να σας πω πως επειδή έχουμε πολλές εκκρεμότητες, σας στηρίζω για όλα όσα έχετε παρουσιάσει. Μπορούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι να χρησιμοποιήσουν ένα λεπτό για τις παρεμβάσεις τους, γιατί έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο και αν ξεκινήσουμε αμέσως, νομίζω θα προλάβουμε. Ο κύριος Στοτοράτσι είναι ο πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ για την προστασία προσωπικών δεδομένων, εσείς προετοιμάζετε την έκθεση για την εφαρμογή της σχετικής νομοθετίας. Εντάξει, στην εφαρμογή θα εξετάσετε και το θέμα των τρόπο με τον οποίο η νομοθεσία αυτή ε, χρησιμοποιείται για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες σε κράτη-μέλη. Επίσης, η ομάδα μας ε, σας έχει στηρίξει από την αρχή για το θέμα της στήριξης του κράτους δικαίου και η Σοφή είπε πολλά. Πιστεύω πως εσείς ε, θα προσπαθήσετε να βοηθήσετε, αλλά δεν ξέρω αν σας στηρίζουν επαρκώ οι υπόλοιποι συνάδελφοί σα στην Επιτροπή. Είδατε τι έγινε με την έκθεση για τη διαφθορά πριν από μερικά χρόνια. Επρόκειτο να έχει και κεφάλαια για κάτι μέλη συγκεκριμένα και μετά ξαφνικά αυτό εξαφανίστηκε και ε, ξεψύχησε. Και μετά ε, το σχέδιο δράση για τη δημοκρατία. Να δούμε και τη σπίδα πει έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα σύμφωνα και με τα λεγόμενά μας. Σκέφτομαι το τι θα γίνει με τη Ρωσία, για παράδειγμα. Έχουμε τα κονδύλια για να καταπολεμήσουμε αυτές τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας. Και νομίζω τα λίγα εκατομμύρια που έχετε προβλέψει δεν είναι αρκετά. Τέλος, κάτι που διάβασε ειδήσει σήμερα. Η νέα πολιτική μετανάστευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν. του Ηνωμένου Βασιλείου, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύουν τα όσα διαβάζουμε, αλλά βλέπω να ε, υποδεικνύονται κάποια στερεότυπα και κάποιες ε, ε, εθνικότητες να κατονομάζονται. Θυμόσαστε τον υδραυλικό από την Πολωνία και τον οικοδόμο από τη Ρουμανία. Πώς θα εξασφαλίσετε πως στους επόμενους μήνες και στις διαπραγματεύσεις οι βασικές αξίες των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ε, τηρηθούν και θα υπερασπιστούν κύριος Ράντιεφ που είναι και ο αντιπρόεδρός μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Γιούροβα, το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία έκθεση για το τι συμβαίνει με τη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία μοναδική έκθεση. Δύο χρόνια αργότερα η επρόκειτο να δημοσιευθεί η δεύτερη έκθεση, αλλά δεν συνέβη αυτό. Και το θέμα της διαφθοράς θεωρήθηκε κομμάτι των όσων συζητάμε στο Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο. Θα είναι κομμάτι λοιπόν του μηχανισμού αυτό για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και τι θα γίνει με την υψηλού επίπεδου διαφθορά, με την κατάχρηση εξουσίας για όσους δεν στηρίζουν το κράτος δικαίου. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συνεχίσει να συντάσσει εκθέσεις για τη διαφθορά. Μήπως χρειαζόμαστε και μια κοινή στρατηγική για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Διαφορετικά δεν θα νομοθετήσετε για ένα θέμα το οποίο είναι ύψης της σημασίας. Η κυρία Πούρεκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, 25 μήνες πέρασαν από τότε που εκκινήθηκε κατά της Πολωνίας η διαδικασία του άρθρου 7. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκτοτε έχει μιλήσει πολύ συχνά για το θέμα του κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς αυτό δεν έχει βελτιώσει την κατάσταση, που έχει χειροτερεύσει κι άλλο, αφού η ε, κυβέρνηση του νόμου και της δικαιοσύνης έχει λάβει κάποιες καταστροφικές αποφάσεις. Είμαι ε, ευρωβουλευτής, είμαι ε, δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρώην επίτροπος για το θέμα αυτό. Θέλω να μου πείτε, εσείς θα βρείτε κάποιο μηχανισμό ο οποίος θα βοηθήσει να εξασφαλίσουμε ε, τον, ε, το κράτος δικαίου έτσι ώστε να μην ε, αισθάνονται τις συνέπειες αυτού οι πολίτες και πότε θα παρουσιάσετε αυτό το σχέδιο δράσης εσείς που είχατε αυτές τις ιδιότητες τις οποίες προανέφερα. Ο κ. Κέρνερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, τρεις ερωτήσεις. Αναφέρατε το μηχανισμό, αυτή την τον ετήσιο κύκλο για, τον, για το κράτος δικαίου. Δεν μπορέσει να το πράξει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Το βλέπετε ως πρόβλημα. Εγώ το βλέπω. Βλέπω μεγάλο πρόβλημα ακόμα και σε επίπεδο αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Και δεύτερον, GDPR, προστασία προσωπικών δεδομένων, τι γίνεται με τις ε, εθνικές αρχές προστασίας, το βλέπω στην Ιρλανδία. Έχουμε προβλήματα εφαρμογής και τρίτον πλατφόρμες, περιεχόμενο, κανόνες. δεν μπορέσετε να πιέσετε λίγο περισσότερο εκεί. Και πώς συγκεράζουμε ελεύθερο λόγο με επιβλαβές περιεχόμενο. Δεν θέλουμε άλλο ένα πόλεμο τύπου Apple και πάλι, χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Ευχαριστώ. Ως εισηγήτρια θέματος, ανησυχώ τα μάλλα σχετικά με τις προτινόμενες μειώσεις του προπολισμού για τα προγράμματα αυτά. Γιατί καλή η τριάδα, καλό το τρίπτυχο των θεμάτων που μας αναφέρατε, αλλά τι γίνεται με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, πώς ακριβώς εσείς ως Επίτροπος μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι κάποια από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες στην Ένωση θα τύχουν προστασίας. Επίσης είστε υπεύθυνοι για την ελευθερία των μέσων. Εμείς γράφουμε σχετικά έκθεση πρωτοβουλίας. Ποιε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε θα αναλάβετε για να προστατεύσετε πιο αποτελεσματικά τους δημοσιογράφους για ειδική νομοθεσία, η ε, οποία κατά των δημοσιογράφων. Εκεί τι κάνετε ειδικά για τις γυναίκες δημοσιογράφους που απειλούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. Τι θα κάνετε για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις παρατηρήσεις της. Κράτος δικαίου και πάλι. Κατάλαβα καλά. Είπατε ότι ευρωπαϊκά κονδύλια τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα υπόκεινται σε κάποιες από τις λεγόμενες αρισιμότητες, σε κάποιες προϋποθέσεις για να καταβληθούν στο κράτο μέλο. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να μην δώσουμε κονδύλια σε κράτο μέλο, εάν δεν περάσει το τεστ. Δεύτερον, η αιτήσια έκθεση που είπατε επί του κράτου δικαίου. Μακάρι να τα πάμε καλύτερα εκεί, σε σύγκριση με τα θέματα διαφθορά. Α, διακόπτη πρόεδρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ στα πολωνικά, χαλική, γιατί η ερώτηση αφορά την Πολωνία και τους Πολωνούς πολίτες, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς. Τρία ερωτήματα. Είναι διάλογος μετά από επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από επίσκεψή σας στην ε, Πολωνία. Ε, ένας Πολωνός πρόεδρος να υπογράφει νόμο που προβλέπει πειθαρχικές διαδικασίες κατά δικαστών. Αυτά είναι τα γεγονότα. Προτίθεστε να στείλετε προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να εφαρμόσει προσωρινά μέτρα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια αυτών των δικαστών. Ποιοι είναι οι κανόνε εν τέλει που ισχύουν όταν 64 δικαστέ διώκονται ήδη και περιμένουν κι άλλοι στην ουρά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιοντσέβα. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Ευχαριστώ. Τονίσετε τη σημασία του κράτους δικαίου. Και ναι, έχουμε μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά τον νέο μηχανισμό. Θα ήθελα όμως να αφιστήσω την προσοχή σας σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, την ελευθερία των μέσων. Χαίρομαι που θεωρείται το θέμα πολύ σοβαρό. Περιμένουμε πολλά όντως από την Κομισιόν προκειμένου. Εγώ τα περισσότερα χρόνια είμαι δημοσιογράφος σε παιδιά μάχης, μια ερευνητική δημοσιογράφος και πρέπει να σας πω από την δική μου πείρα ότι καμία εμπολεμή ζώνη δεν είναι πιο επικίνδυνη από την ερευνητική δημοσιογραφία που έχει να κάνει με την διαφθορά. Χρειαζόμαστε λοιπόν μέτρα για την φυσική προστασία, τη σωματική προστασία των δημοσιογράφων, αλλά και άλλα μέτρα. Σε κάποια κρατημέλη, κυρία Γιούροβα, δημοσιογράφοι δολοφονούνται. Σε άλλες χώρες δεν έχουμε θύματα, όμως ε, το θύμα είναι η δημοσιογραφία. Τα μέσα πολλές φορές είναι βία, σε άλλες περιπτώσεις έχουμε συστηματικά ή μέτρα, σε άλλες περιπτώσεις έχουμε νομοθετικά μέτρα κατά της ελευθερίας των δημοσιογράφων. Λοιπόν, θα καθιερώστε έναν σωστό μηχανισμό παρακολούθησης είναι πολιτική. Θα περιλαμβάνει μόνο η ήπια μέσα μέτρα. Και τι είδου εργαλεία θα προτείνετε συγκεκριμένα υπέρ της ασφάλειας και της ακαιρεότητας, της ομαρικής ακαιρεότητας των δημοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και, και... Κύριε Πρόεδρε, Έχω και εγώ να πω κάτι. ο σας παραπλάνησε. Εδώ μιλάμε για έναν νόμο ο οποίος προβλέπει πειθαρχικά μέτρα, όχι ποινικά μέτρα. Οι δικαστές, οι λογοδικαστέ, είναι άνθρωποι που έδραν τι γυναίκε τους, ε, οδηγούσαν ε, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και υπόκεινται σε ποινικέ διαδικασίε, όχι πειθαρχικέ. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Ας μην συγχαίουμε αυτές τις δύο κατηγορίες και ας μην παραπλανούμε επιτέλου του βουλευτέ. Λοιπόν, κυρία Επίτροπε, δύο ερωτήματα. Πρώτον, μιλάτε πολύ για ισότητα. Τι γίνεται με τους χριστιανούς και τις διακρίσεις κατά των χριστιανών στην Ευρώπη, κατά των χριστιανικών συμβόλων στην Ευρώπη. Είχαμε 3.000 επιθέσεις κατά χριστιανών στην Ευρώπη. Μιλάμε για πέντε επιθέσεις την ημέρα. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, κατά τη διάρκεια των ποριών, των διαδηλώσεων για την ισότητα, είναι ένα σωρό επιθέσεις κατά χριστιανών. Πιστεύω αυτά να περιληφθούν στην ετήσια έκθεση. Και πέρα ότι θα τα αξιολογεί αυτά η Κομισιόν κλπ. Αλλά ποιοι θα είναι οι κανόνες, ποια θα είναι τα κριτήρια Τα έχουμε δει αυτά. Μήπως κάποιοι μη εκλεγμένοι υπάλληλοι θα αξιολογούν τα κρατημέλη εν τέλει. Και τι γίνεται με τις ενεργείες της γαλλικής κυβέρνησης κατά των κίτρων γυλαίκων στο Παρίσι, στη Λιόν κλπ. Ε, και με αυτά παρακαλώ να ασχοληθεί η Κομισιόν, όχι μόνο με τα άλλα. Πρόεδρος, κυρία Βυσνεύσια. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλω να πω ότι και πάλι συζητούμε τεκμερώμενες υποτιθέμενες παραβάσεις του κράτους δικαίου. Στην Πολωνία η εγκληματικότητα μειώνεται, ο κόσμος αισθάνεται πιο ασφαλής και ο κόσμος υποστηρίζει εν τέλει τα μέτρα κατά των συγκεκριμένων δικαστών. Υποτίθεται ότι μιλάμε για κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι πώς θα αξιολογούνται οι σχετικές υποθέσεις. Ο τομέας είναι τεράστιος, δηλαδή θα έχετε και συνομιλίες, είπατε, με εκκλησίες και ούτω καθεξής. Πώς θα εγγυηθείτε την ελευθερία της θρησκείας. Εμεί δεν έχουμε καμία όρεξη να εγκαταλείψουμε, να απεμπολίσουμε τι χριστιανικέ αξίε επί των οποίων οικοδομήθηκε η Ευρώπη. Στη Γαλλία μαθαίνω θέλουν να μετακινήσουν ένα άγαλμα του Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου. Μετά μάθαμε ότι πρόκειται για ψευδοείδηση. Και δυστυχώ αυτέ τι ψευδοειδήσει τι επαναλαμβάνεται. Και το ίδιο κάνετε για άλλε πληροφορίε που αφορούν την Πολωνία. Μετά δεξιοί κατηγορούνται για πράγματα που δεν έχουν κάνει ποτέ. Υιοθετείται λοιπόν την απαράδεκτη ρητορική των αριστερών, απαράδεκτο στην Επιτροπή μας. Δεν υπάρχει διερμηνία από τα γερμανικά. Στα γερμανικά. Στα γερμανικά. Α, στα γερμανικά, με συγχωρείτε. Ναι, με συγχωρείτε. Φαίνεται υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Αλλά δεν υπάρχει διερμηνία ούτε προς τα τσεχικά. Ο κύριος Ρομπέρτη. Κύριε Αντιπρόεδρε, Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Τον Οκτώβριο της περσινής χρονιάς το Κοινοβούλιο ε, και το Συμβούλιο προετοίμασαν μια έκθεση για τους καταγγέλλοντες δημοσίου συμφέροντος και ε, αυτό μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαίου για αδικήματα κατά του δημοσίου συμφέροντος, για οικονομικά εγκλήματα, αδικοπραξίες κλπ. Τι σκέφτεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, μπορέσει να ενταχθεί στις εσωτερικές ένομες τάξεις των κρατών μελών αυτός ο κανονισμός έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα όπως ο διεθνικός, η διεθνική διαφθορά, η διαφθορά που περνάει τα σύνορα. Δεν θα ήταν σκόπιμο να προβλέψουμε έναν κεντρικό οργανισμό ο οποίος να ελέγχει την ε, έγγραψη, ε, την ε, μεταφορά της οδηγίας και την εγγραφή της στο εσωτερικό ένομο δίκαιο, στην εσωτερική ένομη τάξη. Κύριε Ρομπέρτη, νομίζω ότι όλοι λάβατε το λόγο. θα μας απαντήσει η αντιπρόεδρος μας, η Βέρα Γιουρόβα. Εντάξει. Φαίνεται ότι κανένας άλλος δεν θέλει να υποβάλει ερωτήσεις. Η κυρία Γιουρόβα. Άμα μου δώσετε λόγο δεν ξέρω κατά πόσο θα σας τον δώσω πίσω γιατί εθίγησαν πολλά και σημαντικά ζητήματα στα οποία θα ήθελα να απαντήσω. Θα ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις ανά θέμα. Πρώτον, ε, κράτος δικαίου. Ο κύριος Λένερς ε, μίλησε για το κράτος δικαίου και πώς, και πώς μπορούμε να ε, το αποτιμήσουμε μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης αναθεώρησης και αποτίμησης και κατά πόσο το άρθρο 7 έχει βελτιώσει την κατάσταση. Λοιπόν, θα το εντάξω αυτό το θέμα στο ευρύτερο πλαίσιο. Αρχίσαμε να συζητάμε για τη χρήση του άρθρου 7 για την κατάσταση στην Πολωνία το 2017 όταν ε, γινόταν συστηματική παραβίαση του δικαίου από την Πολωνία, όπως είχε αποτιμηθεί από την νομική υπηρεσία μας, αλλά και από τα άλλα θεσμικά όργανα. Το άρθρο 7, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε και τότε εντάχθηκε στη συζήτηση του Συμβουλίου, γιατί θεωρήσαμε ότι η διαδικασία είναι σωστή, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ε, ένας νομικός οργανισμός. Γι' αυτό κρίναμε ότι θα πρέπει να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά και τα κράτη-μέλη, που θα πρέπει να ορίσουν και να ερμηνεύσουν το κράτος δικαίου. Ποιες είναι οι αρχές, ποια είναι τα κριτήρια ποιες είναι οι διαχωριστικές γραμμές που αφορούν τη βελτίωση του δικαστικού τομέα. Και αυτό ήταν και ο στόχος της μεταρρύθμισης στην Πολωνία όταν ξεκίνησε το 2015. Ε, θέλησε η Πολωνία να βελτιώσει το δικαστικό σύστημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδράμει και οικονομικά για κάτι τέτοιο και ενθαρρύνει τη μεταρρύθμιση του δικαστικού πλαισίου και του δικαστικού τομέα, με κατάρτιση δικαστών και ούτω καθεξής. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει τα κράτη-μέλη που βλέπουν τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ μεταρρύθμισης, μεταρρύθμισης που βελτιώνει το πλαίσιο λειτουργίας του δικαστικού τομέα και που γίνεται πολιτικοποίηση του δικαστικού τομέα όπου περιορίζεται η ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής. Και θα πρέπει να πω ότι η συζήτηση στο Συμβούλιο δεν οδήγησε πουθενά. Δεν έγινε ψηφοφορία γιατί δεν υπήρχε επαρκής αριθμός ψήφων. Και φυσικά ε, και εγώ προσωπικά είμαι πολύ απογοητευμένη, αλλά θεωρώ ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 7 είναι σκόπιμη γιατί χρειαζόταν η συζήτηση αυτή. Όταν άρχισα να εργάζομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, θεωρήσαμε ότι μιλάμε για αυτό το τρίπτυχο δημοκρατία, για τη δημοκρατία, ε, για το κράτος δικαίου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ορίζουμε το ε, κράτος δικαίου, έτσι ώστε να μην είναι κανένας υπεράνω του νόμου Δηλαδή το Σύνταγμα περιορίζει τις εξουσίες, δεν τις χορηγεί απλόχερα. Πρέπει όμως ίσως να επενδύσουμε σε μία κοινή κατανόηση αυτού του ορισμού. Τι σημαίνει κράτος δικαίου δηλαδή. Επίσης, μιλήσατε για την ε, αναθεώρηση του κράτους δικαίου, τη μεταρρύθμιση και ποια κριτήρια θα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι κοινωνή εξ αρχής από την προετοιμασία της μεθοδολογίας για την αποτίμηση, διότι το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία του δικαιοδοτικού τομέα, οι ελευθερίες, οι διάφορες ελευθερίες λόγου και εκφράζεστε, όλα αυτά απαιτούν ποιοτική αποτίμηση. Γι' αυτό Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια και ερωτήματα προς τα κράτη-μέλη σε σχέση με την κατάσταση στο κάθε κράτος μέλος και θα ήθελα αυτή η διαδικασία να είναι σαφής εξ αρχής για τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν θα ήθελα στο τέλος του έτους ή τον Οκτώβριο έχουμε την έκθεση περί κράτους δικαίου, όπου κάποιος θα αμφισβητήσει και θα πει ότι εργαστήκαμε με μεροληπτικά στοιχεία. Θα πρέπει να υπάρχουν εγγύησεις. Γι' αυτό και ο συνάδελφος Reinders ζήτησε εμπειρογνώμονες σε μία συνδέσμου για να συνεργαστούμε ως προς τη μεθοδολογία έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να είναι κοινωνή. Αυτό εξήγησα και στην Πολωνία όταν ήμουν στη Βαρσοβία, ότι θα χρησιμοποιήσουμε αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα προσυμφωνηθούν και θα διακρίνονται από διαφάνεια. Αυτό ζητάει και η Πολωνία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Μας λένε η Πολωνία και η Ουγγαρία, μα γιατί εστιάζετε την προσοχή σας σε εμάς. Κοιτάξτε τι κάνουν και άλλοι, γι' αυτό χρειάζεται αυτή η εκτενής αποτίμηση και στο τέλος θα φτάσουμε σε ένα αξιόπιστο απολογισμό για το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη και φυσικά πρόκειται για μία συνταγματική ισορροπία. Αυτό είναι ένα ε, κυρίαρχο θέμα. Αφορά δηλαδή τα κράτη-μέλη. Μιλάμε για μία συνταγματική ισορροπία. Στην έκθεση όμως θα δούμε πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο στα κράτη-μέλη πως ε, υπάρχει προστασία του δικαστικού τομέα κατά της πολιτικοποίησης, κατά της διαφθοράς. Και γι' αυτό η Επιτροπή ε, δεν θα εκδώσει μία μεμονωμένη έκθεση κατά της διαφθοράς. Θα ενταχθεί στην έκθεση περί κράτους δικαίου. Και θα εκδίδουμε αυτή την έκθεση σε αιτήσια βάση. Επίσης θα δούμε ποιες τάσεις καταγράφονται ετησίως, κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και τον πλουραλισμό των μέσων και την ελευθερία του εκφράζεστε στα κράτη-μέλη. Ε, Μία τέτοια εκτενής εργασία δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Μετά λοιπόν από την συνεκτική αυτή έκθεση θα κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε στα κράτη-μέλη ως προς το κράτος δικαίου και ε, αυτό το μέσο θα είναι ένα προληπτικό μέσο εάν υπάρχουν εξελίξεις σε κράτη-μέλη που κινούνται προς μία κατεύθυνση αντίθετη από την επιθυμητή. Αυτό είναι το φιλοσοφικό μας ε, υπόβαθρο ως προς την αναθεώρηση του κράτους δικαίου, της έννοιας αυτής και θέλουμε και την υποστήριξη των κρατών μελών για τη μεθοδολογία. Κάποιος άλλος μου είπε κατά πόσο η, θεωρώ ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν μας υποστηρίζει. Ναι, μετά από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μοραβιέτσκι αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει πλήρης υποστήριξη πλήρης υποστήριξη ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος στις διάφορες χώρες και κατέστησε σαφές ήδη πριν στη δήλωσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτή είναι μία από τις αρχές που είναι αναγκαίες και στις οποίες βασίζεται και επενδύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Ρέντκε με ρώτησε για τη χρήση των κονδυλίων για το κράτος δικαίου, για τις αξίες μας, για τα προγράμματα, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ναι, τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο και στα κράτη-μέλη και αυτή είναι η απάντηση και προς την κυρία Κούνκε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ποτέ δεν θα είναι αρκετά τα κονδύλια και πάντα ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα στο ΕΚΤ, στο πρόγραμμα για τις ε, ευρωπαϊκές αξίες και στο πρόγραμμα Creative Europe και Ψηφιακή Ευρώπη. Αυτές είναι οι πηγές χρηματοδότησης που έχουμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να στηρίξουμε τις προτεραιότητες τις οποίες συζητάμε σήμερα. Θα παρακολουθήσω στενά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν τα προγράμματα αυτά και τα συγκεκριμένα κριτήρια που θα βάλουμε στις προσκλήσεις, γιατί πάντα προσοχή χρειάζεται να δίνει κανείς τις λεπτομέρειες. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε τόσα χρήματα, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνετοί και να επενδύσουμε προσεκτικά στις κατάλληλες δράσεις. Τρομοκρατία. Από όπου και να προέρχεται η τρομοκρατία, είναι κακή και πρέπει να διώκεται. Και βεβαίως οι αρχές επιβολής ε, του νόμου, οι ιδιοκτικές αρχές θα πρέπει να λειτουργούν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ενδυναμώσουμε τη Europol και τη Eurojust με περαιτέρω επιχειρησιακές ικανότητες. Η Europol σε επίπεδο προϋπολογισμού πάει πολύ καλύτερα. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Eurojust. Αλλά επαναλαμβάνω, η Europol θα είναι ισχυρή, με καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, με ασφαλή τρόπο, μεταξύ της Europol και των διοκτικών αρχών όπως επίσης και των υπηρεσιών, μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Για τα ηλεκτρονικά τεκμήρια και την ε, ηλεκτρονική μαρτυρία αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε. Έχει γίνει μια ε, καλή συζήτηση την περασμένη εβδομάδα με την κυρία ε, Ραψίπολα και πιστεύω πως θα πρέπει να επιταχύνουμε τις έρευνες που γίνονται σε διασυνοριακό ε, επίπεδο. Το 85% ε, των αποδεκτικών στοιχείων που χρησιμοποιούν οι εισαγγελίε και οι αστυνομικέ αρχέ είναι σε ψηφιακή μορφή. Τα ψηφιακά δεν γνωρίζουν σύνορα στην Ευρώπη και σύνορα δεν έχει και εγκληματικότητα στην Ευρώπη. Όμως οι αρχές μας έχουν τα σύνορα ε, στα οποία τελειώνουν οι αρμοδιότητες τους, άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορούν να δράσουν και διασυνοριακά. Ελπίζουμε πως θα τελειώσει η νομοθετική ε, διαδικασία για την τρομοκρατία ε, online. Θέλουμε τον, να συνεργαστεί μαζί μας ο κλάδος της τεχνολογίας ε, με σοβαρό τρόπο και όταν αποκαλύπτουν ή ανακαλύπτουν περιεχόμενο ε, τρομοκρατικό να κοινοποιούν τις πληροφορίες αμέσως στις αστυνομίες των κρατών μελών, στις διοκτικές αρχές έτσι ώστε να γνωρίζουμε πως υπάρχει ε, ηλεκτρονικό τρομοκρατικό περιεχόμενο και χρειάζεται κάποιος να αναλάβει δράση αλίπητα γιατί η τρομοκρατία είναι μια πολύ σοβαρή απειλή και θα επαναλάβω δεν εξαρτάται από το αν προέρχεται από τα δεξιά ή από τα αριστερά. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στις αντιδράσεις μας. Κύριε Γιάκη, χαίρομαι που η εγκληματικότητα είναι υπό έλεγχο στην Πολωνία. Εξαιρετικό νέο. Τώρα, για το θέμα αυτό με το πειθαρχικό που θέξατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αμφισβητεί τους διορισμούς των δικαστών. Είναι η εκτελεστική εξουσία ή η νομοθετική η οποία τους διορίζει και στην διαδικασία του άρθρου 7 εμείς εκφράσαμε ανησυχίες για την εμπλοκή τον, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαστικού ε, με ε, μέλη τα οποία διορίζονται από την κυβέρνηση και όχι από τους ομολόγους τους. Αυτό. Γιατί κατά τη γνώμη μας η αναθεώρηση αυτή οδήγησε σε ένα συστημικό πρόβλημα έτσι ώστε υπό το Συντάγμα της Πολωνίας το Συμβούλιο αυτό να είναι υπεύθυνο για την τήρηση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας. Αυτό θέλω να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους της Πολωνίας. Χρειάζεται λοιπόν να επιστρέψουμε στο θέμα και να εξηγήσουμε καλύτερα το γιατί κατά τη γνώμη μας αυτό εμπίπτει στο άρθρο 7. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να γνωρίζουμε πως σε άλλα κράτη-μέλη έχουν δικλείδες ασφαλείας. Για παράδειγμα, η εμπλοκή του δικαστικού στις αποφάσεις. Αυτό σημαίνει στην Αυστρία, Ισπανία, Λετωνία, Τσεχία. Ιρλανδία, Σουηδία. Διάφανες διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ο διορισμός λαμβάνει χώρα, οι ίδιες χώρες. Το δικαίωμα της α, αναθεώρησης της απόφασης να μην διοριστεί κάποιος δικαστής. Αυτό στην Τσεχία και στη Γερμανία. Κύριε Γιάκη, κάνατε συγκεκριμένες ερωτήσεις και προσπάθησα να είμαι πολύ συγκεκριμένη απαντήσεις μου. Να σας πω γενικά πως ποτέ δεν δηλώσαμε πως δεν ε, χρειάζεται πειθαρχική διαδικασία σε κάποιο κράτος μέλος. Αυτό που χρειάζεται είναι να προστατεύσουμε ε, το δικαστικό σώμα έτσι ώστε ε, να κρίνονται σε ποιοτικό επίπεδο και οι αποδόσεις των δικαστών έχουν μια πολύ σημαντική θέση στην κοινωνία οι δικαστές. Αν λοιπόν κάνουν κάτι κακό, και εδώ δεν ε, αναμειγμύω τα ποινικά ή τα ε, πειθαρχικά μέτρα, αλλά αν κάποιος δικαστής σφάλει, θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχική διαδικασία. Το ερώτημα όμως είναι, επί της ουσίας, πώς θα εφαρμόζεται αυτό, γιατί η σχετική ερωτημα ομως ειναι επι της ουσιας πως θα εφαρμοζεται αυτο γιατι τη σχετικη νομοθεσια Ε, συντάχθηκε η εξής πρόταση, το ότι δεν θα πρέπει να απευθύνονται για προδικαστικά ερωτήματα ε, οι, οι δικαστές της Πολωνίας να μην στρέφονται λοιπόν για προδικαστικά ερωτήματα προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Άρα λοιπόν αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ύπαρξη όχι πειθαρχικού κώδικα. Κύριε Τοντορέσκη, ε, κράτος δικαίου, κεφάλαιο κατά της διαφθοράς συγκεκριμένη λίστα με ερωτήσει για τις κρατικές συμβάσεις και προμήθειες και για άλλα θέματα θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε πόσο αποτελεσματική και πόσο εντατική είναι η μάχη κατά της διαφθοράς σε κάθε κράτος μέλος. Κύριε Χαλίτσκι, αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την νομοθεσία που υπεγράφει από τον πρόεδρο Ντούντα και όταν πήγα στη Βαρσοβία είπα είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, υπογράφει ο πρόεδρος τον νόμο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περιμένει την τελική μορφή της νομοθεσίας για να την αξιολογήσει και να αποφασίσει κατά πόσο θα ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση και ποιο θα είναι το πεδίο. Αυτό βρίσκεται λοιπόν ακόμα υπό αξιολόγηση. Ε, Κυρία Κέμπερ. Ε, κατά της διάκρισης ε, της θρησκευτική. Τον κύριο Σχοινά να ρωτήσετε όταν έρθει. Είναι ο υπεύθυνο. Για το διάλογο των εκκλησιών, όπως επίσης και για την ασφάλεια. Εγώ πιστεύω πως όλες οι θρησκείες πρέπει να προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε τα εργαλεία χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε διάκριση και χωρίς να εξαιρούμε οποιονδήποτε. Ίσως όμως να σας δώσει μια πιο ε, εντελεχή απάντηση ο συνάδελφος που είναι αρμόδιος για να προωθήσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Κράτος δικαίου, παύλα, χρήματα στον προϋπολογισμό. Ναι, το έχουμε πει πολύ σοβαρά, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο εργαλείο. Χρειάζεται να υπάρχει κάποια βασική δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο φορολογούμενος πληρώνει και τα χρήματα αυτά μοιράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει βεβαιότητα πως τα χρήματα αυτά προστατεύονται στο κράτος μέλος που τα λαμβάνει δεν μιλώ για τα ταμεία συνοχή, μιλώ για όλα τα κονδύλια. Άρα λοιπόν δεν τιμωρούνται έτσι οι χώρε συνοχής και δεν θεωρώ πως ο κόσμος ο, με συγχωρείτε, ο κανόνας ε, του κράτους δικαίου και ε, των πι είναι το μαγικό ραβδί που ε, θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά μπορεί να έχει αποτρεπτικό ρόλο και αυτό είναι σημαντικό. Και να υπενθυμίσω στα κράτη-μέλη και με τον τρόπο αυτό πως εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου θα πρέπει να εξασφαλίζουν πως το δικαστικό σώμα λειτουργεί, πως η διαφθορά διώκεται, πως οι ε, απάτες στις ε, κρατικές προμήθειες ε, τιμωρούνται. Αυτά είναι τα ελάχιστα που πρέπει να απαιτούμε. Καταθέσαμε μία πρόταση η οποία ήταν αρκετά συγκεκριμένη και έδινε και ένα κατάλογο των σημείων που εκινούν τέτοιου είδους διαδικασίες. Και προτείναμε να έχουμε ε, μία αντιστραμμένη ειδική πλειοψηφία, αντίστροφη ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο για να περάσει το θέμα αυτό. Οι διαδικασίε τώρα και οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό τρέχουν. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ψηφοφορία. Φοβάμαι ότι αν αλλάξουμε την πρόταση αυτή και ζητήσουμε να ε, ψηφίζεται με ειδική πλειοψηφία, θα έχουμε κάτι το οποίο θα λειτουργεί μόνο στο χαρτί. Και δεν ήταν η πρόθεσή μας αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπερασπιστεί στεναρά την αρχική της πρόταση. Το συζητήσαμε σήμερα με τους ε, συναδέλφους επιτρόπους ε, και η γνώμη τους ήταν σαφής. Αυτά λοιπόν. Για την ε, τεχνητή και την προστασία των δεδομένων. Το συζητήσαμε διαμακρών, ειδικά την τεχνητή νοημοσύνη και τη δέσμη μέτρων για τα δεδομένα. Να ξέρετε ότι ό,τι και αν κάνουμε είναι στις προτεραιότητές μας να εγγυηθούμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω GDPR. Διαβάστε τη δέσμη που υιοθετήσαμε σήμερα το πρωί. Θα δείτε πολλές αναφορές στον κανονισμό GDPR. Αφορά και μη προσωπικά δεδομένα, αλλά υπάρχει ένα κεφάλαιο σχετικά με την ανωνυμοποίηση των στοιχείων. Είναι θέμα που και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Εμείς ε, θέλουμε να, να εγγυηθούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εξελίξεων οι κανόνες θα τηρηθούν. Η γενική διαχείριση των δεδομένων είναι υπέρ τη οικονομία, δεν έχει σχέση με το GDPR. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη ω ήπειρο να σημειώσει πρόοδο για το καλό των ανθρώπων, για την οικονομική ευημερία, όχι όμω, επαναλαμβάνω, όχι όμω ει βάρο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό λέει και η δέσμη μέτρων που εγκρίναμε, όπω είπα σήμερα. Ε, επαναλαμβάνω ότι ο κανονισμός GDPR περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ε, είναι έντονα παρόν στο έγγραφο αυτό. Επίσης, τις νέες αυτές εξελίξεις, τον νέο τρόπο σκέψης θα τον ενσωματώσουμε και στην προσεχή αναθεώρηση του κανονισμού GDPR. Αυτό τον Μάιο πια Θα εξετάσουμε όλα όσα αναφέρεται. Δεν είναι μόνο ο κανονισμός GDPR εν της νέας στρατηγικής. Ε, το θέμα είναι και πώς λειτουργεί και τι επιπτώσεις έχει ο GDPR στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε επίσης ο κανονισμός να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου και αυτό θα το ξαναδούμε. Θέλουμε να εγγυηθούμε την αρχή μία ήπειρος, μία νομοθεσία. Και αυτό για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής. Να προστατεύεται η ιδιωτικότητα λοιπόν των ανθρώπων σε όλη τη χώρα και με τον ίδιο τρόπο, να μην είναι ακριβή σε κάποια χώρα και φτηνή αλλού. Και ο κύριος Τεντοράτσα ρώτησε κάτι συναφές. Όντως, εξετάζουμε τις περιπτώσεις που ο κανονισμός GDPR χρησιμοποιείται για τον λάθος σκοπό για να περιορίσει για παράδειγμα την προσβεστή πληροφορία. Σε κάποιε χώρες ο κανονισμός είναι αντικείμενο εκμετάλλευση κατά των δημοσιογράφων για να τους περιορίσει. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε πότε και πώς ισχύει ο GDPR να εφαρμόζεται με τον σωστό τρόπο. Το συζήτησα και αυτόν με τον Μάρκ Ζούκερμπερκ πριν από λίγες μέρες. Ζήτησα δεδομένα για την έρευνά μας για να ξέρουμε τι συμβαίνει στα περίφημα μαύρα κουτιά, στους αλγορίθμους αυτούς, βάσει των οποίων γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων των πολιτών μας. Τι γίνεται με τα κηρύγματα μίσους, ποιοι είναι πίσω από αυτά τα κηρύγματα, δεν έχουμε στοιχεία. Οι δικηγόροι από την άλλη μεριά φοβούνται τον GDPR, πολύ ωραία, να το δούμε, να δούμε πώς θα διευκρινίσουμε περαιτέρω αποσαφηνίσουμε ότι ο κανονισμός δεν έχει στόχο να αποτρέπει τους ενδιαφερμένους από το να δίνουν πληροφορίες, στοιχεία στους ερευνητές. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θα τα δούμε σε σχέση με τον κανονισμό GDPR. Τα είπα βεβαίω στην εισαγωγή μου. Δεν σκοπεύουμε να αναθεωρήσουμε τον GDPR, όμως θα εξετάσουμε θέματα εφαρμογή και επιβολής. Για τα θέματα λειτουργία του Ιρλανδικού, της ελληνικής Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, ξέρω την υποπίεση, διότι πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν την έδρα τους στην Ιρλανδία, εκεί έχουν τα κεντρικά τους γραφεία. Είμαι σε επαφή με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιρλανδίας για να διασφαλίσουμε ότι έχουν τις δυνατότητες που χρειάζονται. Αν όχι, κάτι πρέπει να κάνουν να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους. Τώρα, γενικώ οι ικανότητες και οι δυνατότητες αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης. Ρωτήσατε αν είμαστε εξοπλισμένοι οικονομικά για την αντιμετώπιση, τον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης. Η Stratcom έχει αυξημένο προϋπολισμό πλέον. Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τον προϋπολισμό Υπουργείων όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας. Ζητήσαμε από τις ε, φορολογικές αρχές να αυξήσουν, να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να εντοπίζουν επιβλαβές περιεχόμενο, να βεβαιωθούν ότι μπορούν να το αποσύρουν, να το κατεβάζουν, όταν είναι δηλαδή ε, παράνομα οι επιβλαβές, όπως στην περίπτωση συγκεκριμένα της παραπληροφόρησης. Θα συνεχίσουμε επίσης να συλλέγουμε περισσότερα στοιχεία, περισσότερα δεδομένα, περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο δράσης, για την προστασία της δημοκρατίας που θα δημοσιεύσουμε πέρι τα τέλη του έτους, όπως προείπα. Ο αγώνας κατά της παραπληροφόρησης, ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Η προστασία των εκλογών επίσης, η προστασία της ανεξαρτησίας της δημοσιογραφίας. Αυτά βεβαίω αλληλοσυνδέονται. Και με ρωτήσετε αν θα λάβουμε μόνο ήπια μέτρα ή πιο συγκεκριμένα με τη μορφή νομοθετικών ρυθμίσεων. Στον τομέα της εκλογικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών κομμάτων, εκεί που έχουμε αρμοδιότητα, θα εξετάσουμε την διαφάνεια της χρηματοδότησης των κομμάτων Επίσης, κατά αναλογία θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τις πιο κρίσιμε περιόδους πριν από τις εκλογέ. Ξέρετε, έχουμε πολύ καλούς κανόνες για τις εκτός διαδικτύου εκστρατείες, αλλά στο διαδίκτυο δεν πάμε και τόσο πολύ καλά. Χρειαζόμαστε καλύτερους, πιο αποτελεσματικούς κανόνες. Επίσης, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να θεσπίσουμε νομοθεσία για την παραπληροφόρηση. Όμως θα έτεινα να πω, με μια προσωπική άποψη αυτό, ότι εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην ε, φτάσουμε στο άλλο άκρο, στην λογοκρισία. <laughs> Η λογοκρισία δεν ταιριάζει στην Ευρώπη. Και ε, είμαι επίσης κατά της ανάδειξης των φορολογικών αρχών σε κριτές της αλήθειας. Αυτό δεν γίνεται. Διότι αν τελικά δεν θέλουμε να σύρουμε μια διαχωριστική ε, γραμμή μεταξύ αλήθειας και ψεύδους, το να καταφύγουμε στον Μάρκ Ζούκερπερ, για παράδειγμα, στους γίγαντες είναι παραλογισμός. Αυτό όχι, δεν είναι μέρος του σχεδίου μας. Αυτό που μπορεί να δείτε στην πρότασή μας είναι να εντείνουμε τις εργασίε μας για να γίνουμε πιο ανθεκτικοί στην παραπληροφόρηση με βάση τα πραγματικά περιστατικά, με βάση αριθμητικά στοιχεία, με βάση την εμφάνιση των ψευδοειδήσεων στο διαδίκτυο. Θα έχουμε εκτεναμένε διαβουλεύσει μεγάλες διάρκεια για όλα αυτά, γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Επίση θα δράσουμε κατά των κηρύγματων μίσου. Δεν θέλω να δώσω μεθυμένες σε κανένα, αλλά ως δικηγόρος θέλω να το επαναλάβω. Η παιδική πορνογραφία, η τρομοκρατία, κάποια κλεψίτυπα, καταναλωτικά προϊόντα, οι ψευδοειδήσεις, όλα αυτά είναι απαγορευμένο περιεχόμενο, το οποίο δεν θέλουμε να βλέπουμε στο διαδίκτυο, ούτε εκτός διαδικτύου βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο στην νομοθεσία περί της ψηφιακής αγοράς. Θα απαγορεύουμε αυτό το παρανομό απαγορεύεται ούτως ή άλλως αυτό το περιεχόμενο, αλλά στο δικό μας σχέδιο δράση, τη δημοκρατία, θα αναφερόμαστε και σε περιεχόμενο το οποίο δεν είναι ε, αναγκαστικά παράνομο, αλλά είναι επιβλαβές. Κύριε Γυρόβα, εσείς μου είπατε ότι θα σταματήσετε κάποια στιγμή να πάρουμε τον λόγο. Πείτε μου πότε. Πρόεδρος, Βλέπω κάποιες αντιδράσεις από αυτούς που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν ή δεν ξέρω αν κάποιοι θέλουν να επανέλθουν για δευτερολογία. Κύριε Μπάρλε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Έστειλα μια γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν στις 6 Ιανουαρίου. Δεν έχω πάρει έκτορη απάντηση. Οπότε, με την ευκαιρία, να ρωτήσω αν όλοι συμφωνούμε μετά και από τις αποφάσεις, ε, τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να ρίξουμε μια ματιά στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και καλό είναι να βλέπουμε την γενικότερη εικόνα, έτσι. Με βάση λοιπόν αυτά, πώς θα προχωρήσετε σε δράση για όλα αυτά μαζί. Δηλαδή, Πώς θα έχουμε αποτελεσματικό έλεγχο, εάν το κρατός κατά πρώτο λόγο σας υποδεικνύει ποιες είναι οι πηγές των στοιχείων. Στην περίπτωση τώρα της προνοίας, θα συμφωνούσατε ότι αυτή η τελευταία μεταρρύθμιση αποτελεί μια διάσταση στον αγώνα που γίνεται κατά του κρατούς δικαίου, έτσι όπως το βλέπουμε στην Ευρώπη. Μήπως κινδυνεύουμε να χάσουμε το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, εργαλείο εφαρμογής του κρατούς δικαίου. Σοφία Βέλτ, αλλά πάρα πολύ γρήγορα γιατί... Ε, δεν ξέρω αν έχασα την απάντηση, αλλά ο Σάλφος ο Τράγος ε, είπε ή μάλλον ρώτησε αν θα έχουμε συστάσεις ε, αναχώρα μετά την πρώτη έκθεση. Και εγώ δεν ξέρω να το άκουσα αυτό. Ναι, τι γίνεται με την κατάσταση με τους ε, προσωρινούς εισαγγελείς. Ωραία κύριε Γύροβα, έχετε δύο λεπτά για να απαντήσετε και σε αυτά. Για την Πολωνία μια νέα διάσταση. Δεν ξέρω, αποτελεί μάλλον συνέχεια της ε, μεταρρύθμισης. Η Κομισιόν θα το εξετάσει όπως έκανε και στο παρελθόν. Θα αξιολογήσουμε τη νέα κατάσταση και θα προχωρήσουμε ένα λόγο αν... Με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου, λέει ο Ιταλός βουλευτής. Ναι, Με συγχωρείτε, λέει η Επίτροπος. Πήρα τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά. Οπότε, συνεχίζω. Λοιπόν, έχουμε ως Κομισιόν τα παραδοσιακά εργαλεία για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. για τον, με για τον ε, ευρωπαϊκό Συγγελέα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με προσωρινούς διορισμούς. Ούτε μπορούμε να έχουμε εισαγγελείς. 50% για την εσωτερική νομή τάξη και 50% για τον ΕΠΠΟ. Αλλά εντάξει, αν το θέλει το κράτο μέλο, ίσω. Ε, νομίζω ότι θα είναι εξίσου επαγγελματίε. Όταν μιλήσαμε για τον Ευρωπαίο εισαγγελέα, ε, είχα πει ότι χρειαζόμαστε τους καλύτερους τους αρίστους για τη θέση αυτή. Για το επιτελείο του Ευρωπαίου εισαγγελέα, γιατί θα αντιμετώπιζε υποθέσεις, ας πούμε, μεγάλης πολυπλοκότητας οικονομικού εγκλήματος. Εκεί, όπως είπα, θέλουμε τους ε, καλύτερους και υποστήριξα τον αρμόδιο επιτροπό. Πρέπει να βοηθήσουμε την εισαγγελέα. Είναι υποχρέωση της Κομισιόν να το πράξει αυτό, να αναμαζέψει λέει, τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω της. Σε σχέση με τον μηχανισμό ελέγχου των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης, Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουμε τις συστάσεις ε, των κρατών. Θα έχουμε εκθέσεις αναχώρα, θα έχουμε και το επίπεδο συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών και θα ολοκληρώσουμε με την αποτίμηση της κατάστασης στα κράτη-μέλη, αλλά δεν θα ακολουθήσει την ίδια μορφή με αυτή του ε, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ναι, χώρα προς χώρα. Τα κράτη-μέλη έχουν δύο για να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία. Για ορισμένα κράτη-μέλη χρειάζεται περισσότερη εργασία γιατί ε, σε σχέση με αυτούς τους ε, καταλόγους που καταρτήσαμε χρησιμοποιήσαμε ορισμένα παραδείγματα από κράτη-μέλη για να ορίσουμε διαφορετικούς ε, διάβλους, διάβλους επικοινωνίας και διάβλους ενημέρωσης. Θα σας βοηθήσω όσο το περισσότερο μπορώ αν δω ότι υπάρχουν κράτη που έχουν μείνει πίσω μέχρι την πλήρη εφαρμογή σε σχέση με την οδηγία για τους καταγγέλλοντες δημοσίου συμφέροντος. Δεν ήταν εύκολο να εφαρμοστεί, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί, αλλά θεωρήσαμε ότι πρέπει να έχουμε νομοθεσία σε όλα τα κρατημέλη. Σε σχέση με τον έλεγχο των μέσων, στις 18 Μαρτίου θα ε, δημοσιεύσουμε το, τη νέα κατάσταση πλουραλισμού των μέσων σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στα κράτη-μέλη, νομοθεσία, ασφάλεια, ε, νομικά ζητήματα τις πολιτικές πιέσεις στα τοπικά μέσα, τις οικονομικές πιέσεις εις βάρος τους και την αρχή του μη αποκλεισμού και θα γίνει και μια διάσκεψη για τα μέσα στις 20 Μαρτίου όπου θα συνεργαστούμε με κάθε κράτος μέλος χωριστά γιατί θα έχουμε έναν απολογισμό αναχώρα το Μάιο-Ιούνιο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιουρόβα. Προσπαθήσατε να δείτε διεξοδικά όλα τα θέματα μέσα σε μια μισή ώρα. Θα σας ξαναδούμε και θα σας ξανακούσουμε με το πέρασμα του χρόνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Χινάς, περιμένει ένα λεπτό μέχρι να επαναλάβουμε τις εργασίες μας. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Σχοινά, που είναι εδώ μαζί μας. Χωρίς καθυστέρηση είχαμε τον πρώτο διαρθρωμένο διάλογο, τον πρώτο γύρο πριν τώρα ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Χινάς, που προωθεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, θα μας μιλήσει για συναφή θέματα και θα μας μιλήσει ιδιαίτερα για την ολοκλήρωση της Ένωσης Ασφάλειας και την αντιμετώπιση παραδοσιακών και συγχρόνων απειλών. Λοιπόν, θα έχουμε τον πρώτο γύρο συντονιστών που θα μιλήσουν για δύο λεπτά έκαστος ε, και τα μέλη επίσης θα μπορέσουν να εκφραστούν στη συνέχεια για ένα λεπτό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαστε εδώ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Η αίθουσα αυτή μου φέρνει πολλές μνήμες. Στις 3 Οκτωβρίου έγινε η ακροασή μου και σας είπα τότε ότι θα με βλέπετε πολύ συχνά. Να λοιπόν που είμαι εδώ ενώπιόν σας για δεύτερη φορά από τότε που αρχίσαμε τις εργασίες μας στις 2 Δεκεμβρίου. Σήμερα θα σας μιλήσω για το άλλο μωρό της οικογένειάς μου που είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια της Ένωσης. Σήμερα το πρωί είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την εφαρμογή του Δουβλίνου σήμερα το πρωί. Πολύ σημαντικό θέμα και αν θέλετε μπορούμε να το θίξουμε εν μέρη γιατί ήταν το κέντρο βαρύτητας των συζητήσεών μας ε, όταν βρεθήκαμε στο Στρασβούργο. Για την ασφάλεια της Ένωσης είχαμε πει ότι θα πρέπει να δούμε τις παραδοσιακές και σύγχρονες απειλές και θα θέλαμε η Ένωσή μας να μπορέσει να αποδώσει και να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς στους δρόμους και στα σπίτια τους και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός και εμένω αυτή τη δέσμευση. Ο Σερ Τζούλιαν Κίνγκ ήταν ο πρώτος επίτροπος στην προηγούμενη επιτροπή που όρισε αυτό το νέο σύστημα ασφάλειας, ε, αυτό το νέο γαλαξία με τους διάφορους πλανήτες και αποτελεί επιτυχία για την Επιτροπή, ώστε να μην υπάρχει ο κατακαιρματισμός που υφίσταται μέχρι τούδε με τους διάφορους πέκτες και τη στρωματοποίηση ασφάλειας που υπήρχε μέχρι τώρα. Μιλάμε λοιπόν για μια στρατηγική για την ασφάλεια της Ένωσης και το επόμενο επίσημο βήμα θα γίνει τον Ιούνιο πριν από το καλοκαίρι όπου θα παρουσιάσουμε μία νέα συνεκτική στρατηγική για την ασφάλεια στην Ευρώπη που θα χαρτογραφήσει τη δραστηριότητά μας για την επόμενη πενταετία. Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς βασιζόμαστε σε τέσσερα μπλοκ, την ε, ε, διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία και ανταλλαγές πληροφοριών, αντιτρομοκρατία και έλλειψη ριζοσπαστικοποίησης, οργανωμένο έγκλημα και ασφάλεια στην ψηφιακή εποχή, καθώς και νέα ζητήματα όπως την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την, ε, την ε, υβριδική ασφάλεια και την διάρθρωση στον ψηφιακό τομέα. Όπως και στο παρελθόν θα συνεργαστούμε και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εργασία σας καθώς και την Επιτροπή κατά της ε, τρομοκρατίας, την Επιτροπή ΤΕΡ. Ας, ας κάνουμε μία ομαδοποίηση θεμάτων. Καταρχήν την συνεργασία αστυνομικών αρχών ε, και ανταλλαγή πληροφοριών διασυνοριακά, έτσι ώστε να κλείσουμε το χάσμα πληροφοριών για να εξασφαλίσουμε την εσωτερική ασφάλεια. Προετοιμάζουμε διάφορες πρωτοβουλίες σε αυτό το τομέα. Στο πρόγραμμα εργασίας φέτος θα προτείνουμε προτείνουμε μία στοχοθετημένη αναθεώρηση του κανονισμού της Europol, έτσι ώστε η Europol να γνωρίζει πολύ καλά και να ενημερώνεται για τα εγκλήματα και την εμβέλειά τους μέσα στα πλαίσια της νέας εντολής των κρατών μελών για τις απειλές ασφάλειας. Επίσης, να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός ε, της Europol με τον κανονισμό EDPS για να μπορέσουμε να ε, προστατεύουμε καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, ανταλλαγή πληροφοριών διασυνοριακά και εδώ μιλώ για την διαλειτουργικότητα συστημάτων πληροφοριών, αιτίας, ΙΕΣ και άλλων και γνωρίζω ότι μιλάμε για συγκεκριμένα μέσα για να αυξήσουμε την ικανότητά μας να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να μπορούν οι επικεφαλείς να ανταλλάσσουν πληροφορίες εν ευθέτω χρόνο. Ο Ζωζέ Μπορέλ ε, θέλει να ε, ενισχύσει τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, με στρατηγικές χώρες και γειτονικές χώρες ως προς τα χάσματα πληροφορίας και για πρόληψη, ανείχνευση και έρευνα ως προς, εγκλήματα, ως προς σοβαρά εγκλήματα και τρομοκρατία. Ως προς την τρομοκρατία και την πρόληψη ρίζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε εξτρεμισμούς, εδώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε την κοινωνική σύνοχη και να δούμε τις ρίζες της κακοδαιμονίας που ε, δημιουργούν και οδηγούν σε αυτή τη βία. Νομίζω ότι θα συζητήσατε με την κυρία Γιούροβα τα δικά της, τη δική της πτυχή του θέματος, αλλά μιλάμε για εξτρεμισμό και τρομοκρατία που αποτελούν απειλή ασφάλειας και άμεση απειλή για την ειρηνική συνύπαρξη της, ε, κοινότητας, της κοινότητάς μας. Γι' αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και με σφαιρικό τρόπο. Στο παρελθόν έχουμε διευρύνει τη στήριξη όχι μόνο προς τους ε, ε, πραγματογνώμονες και τους όσους στην πράξη επιχειρούν, αλλά και σε όσους βρίσκονται στις ε, ε, γειτονικέ μας χώρες και να σας πω πως έχουμε περιχαρακώσει 60 εκατομμύρια ευρώ ε, για τους ερευνητές, για όσους χαράσουν πολιτική και για όσους επιχειρούν, έτσι ώστε να καταφέρουμε μια πραγματική ε, παρέμβαση στα όσα συμβαίνουν. Και έχουμε και ένα κλάστερ ακόμα ε, που είναι αυτό, η συμφωνία για το τρομοκρατικό περιεχόμενο online είναι κάπως απογοητευτικό που παρόλα τα όσα συνέβησαν στο Christchurch και σε άλλες περιοχές και σε παρόμοια γεγονότα δεν καταφέραμε σε θεσμικό επίπεδο να βρούμε μια συνολική συμφωνία η οποία θα μας επέτρεπε να περάσουμε σε μια διασυνοριακή, σε εντάλματα διασυνοριακά ε, επίγουσας απόσυρσης τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. Αντίθετα, χρησιμοποιείται το ε, περιεχόμενο αυτό για να ριζοσπαστικοποιήσει ε, πολίτες και δεν ε, προλαβαίνουμε να παρέμβουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αυτοματοποιημένα εργαλεία. Δηλαδή, 50 χρόνια θα χρειαστούν τα γραφεία στα οποία αναφέρονται αυτές οι παραβιάσεις, εάν χρειάζονταν να εξυπηρετήσουν όλες τις αναφορές που λαμβάνουν. 1,5 ε, εκατομμύρια φορές χρειάστηκε να παρέμβει η Google για να αφαιρέσει οι ε, εικόνες από την επίθεση στο Christchurch. Οπότε δεν μπορεί να γίνεται πια με ανθρώπινο χέρι, πρέπει να γίνεται αυτοματοποιημένα. Και επειδή ε, πλησιάζει η επέτειος των γεγονότων στο Christchurch, ελπίζω πως μπορείτε να με βοηθήσετε για να φέρουμε αυτή την προσπάθεια ε, σε πέρας. Να σας πω λοιπόν ε, καταρχήν για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο πως είναι ένας πλανήτης που γίνεται όλο και πιο κοντινός γιατί η τεχνολογική πρόοδος έχει επηρεάσει το πώς ε, επηρεάζει το οργανωμένο έγκλημα τη ζωή μας και στο κυβερνοχώρο θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους, τα παιδιά, όσους πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, με στοχευμένες προτάσεις, οι οποίες θα φέρουν ένα αποφασιστικό χτύπημα με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά ε, την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών με συγκεκριμένα στοιχεία για μια ε, δραστήρια και ε, στεναρή απόκριση που θα συνδυάζουμε τις προσπάθειες που κάνουν στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα για να προστατεύσουμε όλοι μαζί τα παιδιά μας τέλος, στην πολιτική ε, ασφάλειας για την ψηφιακή εποχή, η οποία συζητιέται αυτή τη στιγμή, γιατί σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το ψηφιακό πακέτο. Είναι μια πρώτη προσπάθεια να πλησιώσουμε ένα εξαιρετικά περίπλοκο θέμα που είναι ο τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία μας και το πώς μεταχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πιστεύω πως η προσέγγιση μας στην ασφάλεια και στην προστασία δεδομένων των ε, εξελίξεων θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και online και offline. Δεν έχουμε χρόνο ε, και περιθώριο ε, για, τις, ε, για να προλάβουμε τις τεχνολογίες αυτές και κυρίως δεν θα διαδοθούν αν δεν εξασφαλίσουμε πως είναι ασφαλής για όλους. Την περασμένη μήνα παρουσιάσαμε ε, μία χρηστή προσέγγιση για την τεχνολογία του 5G με έναν τρόπο που θα μας εξασφαλίσει και θα μας βοηθήσει. Είναι καταπληκτική τεχνολογία η οποία όμως δεν μπορεί να ε, εξαπλωθεί εις βάρος της ε, εσωτερικής ενιαίας αγοράς. Θα δούμε πώς μπορούμε να λάβουμε την και να ακούσουμε την άποψη όλων των εμπλεκομένων που δεν είναι οι συνήθεις, οι υποπτοί, όχι αυτοί που γνωρίζουν τα θέματα και είναι ε, πρόθυμοι, αλλά οι πολίτες. Να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους πολίτες μας, από τις κοινωνίες μας, για να γίνει μια πλούσια συζήτηση 20 εκατομμύρια ευρώ για την ε, τεχνητή νοημοσύνη και την έρευνα για το πώς αφορά τις ε, διοκτικές αρχές και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτές, έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τι προσφέρουν αυτές τις τεχνολογίες. Τα επόμενα χρόνια πρέπει να καταλάβετε πως εκτός από φίλους και οικογένειες θα έχουμε και ε, κάποιους φιλικούς εχθρούς ή εχθρικούς φίλους έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη και αυτή είναι αυτός ο κίνδυνος που θα χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη να είναι ευρωπαϊκή. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και είναι ένας χώρος στον οποίο η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να δράσει τώρα να κάνει τα δύο που ξέρει να κάνει καλά η Ευρώπη. Καταρχήν, ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο και δεύτερον αυτό να το κλιμακώσει μια και είμαστε μια μεγάλη αγορά την οποία δεν μπορεί κανείς να αγνοεί ε, να την αγνοούν ούτε οι ε, διαταράκτες, ούτε αυτοί οι οποίοι απειλούν τις αξίες και τις αρχές μας. Να κλείσω λοιπόν με ένα πολύ σημαντικό σημείο. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω και έχω αναφερθεί προηγουμένως και στην ακρόασή μου, αλλά ε, χαίρομαι που μπορώ να τα επαναλάβω. Καταρχήν, κάθε μία από τις προτάσεις μας για την Ένωση Ασφάλειας θα σχεδιάζει και θα εντάσσει την πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι δική μου προσωπική δέσμευση, προσωπική μου προτεραιότητα. Είπα ότι δεν θα το κάνουμε έτσι, λίγο στο παραπέντε. Θα είναι μια, ένα προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε με την ε, ένωση αυτή. Και το δεύτερο, που είναι ένα αγαθό απαραίτητο για να έχουμε αυτή τη μεγαλύτερη αγορά ασφάλειας, ε, ένωση ασφάλειας, με συγχωρείτε, είναι η εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και δομές ασφαλείας δεν εμπιστεύονται κανέναν. Αυτή είναι η νοοτροπία τους. Και για να είναι αποτελεσματικοί λένε και να προστατεύουν την ασφάλεια δεν θα πρέπει να εμπιστεύεστε κανέναν. Αυτό δεν είναι αρκετά καλό για όσα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη σε επίπεδο θεσμών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δείξουμε πως δεν θα φέρουμε επικαλύψεις με ό,τι έχουν κάνει αλλού στην κοινωνία μας και θα πρέπει να αποδείξουμε στην κοινωνία πως η ευρωπαϊκή δράση προσφέρει ε, προσθέμενη αξία είναι ένας καταλήτης που βελτιώνει τα όσα γίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, όπως και προηγουμένως θα συζητήσουμε τρώντας το χρόνο. Έχουμε χρόνο ως τις 6. Έχουμε μία ώρα και κάτι, αλλά δεν έχουμε μόνο τους συντονιστές, τον πρώτο γύρο. Έχουμε και όλους τους άλλους, οπότε συντονιστές δύο λεπτά μόνο παρακαλώ, κάντε ό,τι μπορείτε, ώστε να μιλήσουν στη συνέχεια όσο δυνατόν περισσότεροι βουλευτές. Κύριε Λένα, παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Σχοινά. φαντάζομαι ήταν πολύ εξαντλητικό να ταξιδέψει όλε όλες τις ε, πρωτεύουσες. Χαίρομαι που είστε εδώ ε, για να συζητήσουμε και το άλλο μωρό σας, όπως είπατε και εσείς. Αλλά έχουμε δύο μωρά, μην το ξεχνάμε αυτό. Μια νέα ναυτική αποστολή στην Μεσόγειο, η οποία θα εκκραστήσει την Σοφία. Είπε ότι... Ο είπε ότι θα αποσυρθούν εν καιρό και όταν ε, δεν υπάρχουν πλέον αποδείξεις παράνομης διακίνησης. Λοιπόν, πώς θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Και δεύτερον, υπογραμμίσατε την σημασία της λειτουργικής συμβατότητας των συστημάτων πληροφοριών μας. Δεν το κάναμε την προηγούμενη φορά. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά σε επίπεδο μέλους. 16 κράτη-μέλη δεν έχουν εθνικό σχέδιο εφαρμογή. Καταλαβαίνετε ότι είναι υπερβολικά ίσω φιλόδοξο το έργο αυτό, οπότε παρακαλώ πιέστε αυτά τα κράτη-μέλη και ενημερώστε του υπολείπου. Α, και ένα τρίτο, συγγνώμη, θα είμαι σύντομο. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνεδρίο αξιολογεί τα αισθήματα πληροφοριών, τι είναι με τα δεκτυλικά αποτυπώματα, ναι, μόνο 10 κράτη Σέγγεν είναι έτοιμα να χρησιμοποιήσουν τις νέες λειτουργικές δυνατότητες. Μετά άλλα κράτη-μέλη παραπονούνται ότι παίρνουν περιβολικά πολλές πληροφορίες από αναζητήσεις με βάση αλφαριθμητικά στοιχεία, έχουν πολλά ε, πλάστα ε, θετικά. Συμβαίνει αυτό σε περιβολικά υψηλό ποσοστό των αναζητήσεων Απαραίτητα υψηλό ποσοστό. Τι κάνουμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και τέλος για το 5G. Είπατε, ορθώς πιστεύω, υπάρχουν ερωτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των διασυνδέσεων με συσκευέ. Εγώ έχω και άλλες ερωτήσεις σχετικά με την αστυνομία, τα σώματα ασφαλείας, ε, κάποια συστήματα που λειτουργούν στο 4G, στο 4G μπορεί να μην λειτουργούν στο 5. Ε, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα σώματα ασφαλείας θα συνεχίσουν να είναι σε θέση να φέρουν σε πέρα τις αποστολές τους επί 5G όπως και επί 4G. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο σχεδόν κάλυψε ήδη ο συνάδελφος. Ξέρετε, θεσπίζουμε ένα σωρό μέτρα και κανόνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και μετά δεν βλέπουμε εφαρμογή. Και δεν άκουσα πολλά γι' αυτό το θέμα η λειτουργική συμβατότητα ήδη ανακοινώθηκε, θα χρειαστεί χρόνια γι' αυτό, κάποια κρατημέλη έχουν καν ξεκινήσει και να αναφέρω και ένα παλιό μέτρο πριν, το οποίο ούτε αυτό εφαρμόστηκε. Λοιπόν, πώς θα βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση, τη μη εφαρμογή τέλο πάντων. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να ανακοινώνουμε μέτρα και μετά να μην εφαρμόζουμε τίποτα. Αν δεν εφαρμόσουμε τίποτα, δεν έχει κανένα νόημα να ψάχνουμε που, που βάζουν νερό κάποιοι νόμοι. Μετά συνεργασία αστυνομία με δικαστική εξουσία, αυτό μπορεί να γίνει μόνο επιγραμμικά, μόνο διαδικτυακά. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερες κοινέ ομάδε έρευνα σε ειδικέ περιπτώσει εγκλημάτων, για ειδικέ μορφέ εγκληματικότητα, εκεί που οι εμπειρογνωμονε θα δρουν από κοινού ταχύτερα για να μπορούν ε, από κοινού πρώτα απ' όλα να λαμβάνουν αποφάσει, να έχουμε εντωμεταξύ καλλιεργήσει η εμπιστοσύνη μεταξύ των ομάδων και ούτω καθεξή. Όσον αφορά σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση παιδιών κλπ. Πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι επικεντρωνόμαστε περιβολικά στο επιγραμμικό κομμάτι, στο διαδίκτυο, αλλά το θέμα είναι αυτές τις προσπάθειες να τις συνδυάσουμε αυτές που γίνονται στην πράξη. Στην πραγματική <laughs> πραγματικότητα δηλαδή. Γιατί οι άνθρωποι που είναι στο διαδίκτυο δραστηριοποιούνται και στον πραγματικό κόσμο, ξέρετε. Πώς θα γίνουμε λοιπόν καλύτεροι, πώς θα ενημερώσουμε, πώς θα ευαισθητοποιήσουμε για να πιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και τέλος, έχετε μια ιδέα για το τι θα κάνουμε για το εξή θέμα. Όσο όλο και περισσότερα παιδιά δέχονται μηνύματα, προσκλήσεις από ανηλίκους στο διαδίκτυο που, τους, που τα προσκαλούν, ε, τα καλούν να κάνουν πράγματα μπροστά στην ε, κάμερα του υπολογιστή, πράγματα που ένα παιδί δεν θα έπρεπε να κάνει. Είναι και αυτό κάτι περί του οποίου πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε τα παιδιά και το περιβάλλον τους. Και εδώ είπα και ξαναλέω, χρειάζεται οι οργανώσεις γονέων να μιλήσουν, οι γονείς οι ίδιοι να μιλήσουν στα παιδιά, να τα ενισχύσουν έτσι ώστε να μπορούν να αντιδρούν. Και η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Αναφέρεται θέματα όπως το δίκτυο RAN, το θέμα της συνοχής των δρασιών μας, αλλά πιο συγκεκριμένα. Τι δράσεις έχετε προκρίνει, με ποια κονδύλια. Μιλώ για πραγματικά μέτρα. Και ξέρετε, στο πεδίο, όπω λέμε, οι χώρε διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι αιτίε που οδηγούν στην ριζοσπαστικοποίηση είναι διαφορετικέ από χώρα σε χώρα. Αν δεν κάνω λάθο, κάτι είχα πει για δύο λεπτά, αλλά Κύριε Εντεβέλτ. Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Καλώς ήλθατε, Επίτροπε. Για την ομοθέτηση νόμων. Είπατε να κάνουμε γρήγορα πράγματα για τα τρομοκρατικά μηνύματα στο διαδίκτυο. Ναι, σύμφωνοι. Σπέβδε βραδέ όμω γιατί βραδέως όμως πρέπει να κινηθούμε σωστά. Η Κομισιόν μας ε, λέει συνεχώς πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, βιαζόμαστε και όταν έρθει η στιγμή να πάμε παρακάτω και τα στυλώνει το Συμβούλιο, εκεί ε, δεν ε, τους λέμε πιο γρήγορα, απλώς αποσύρουμε τις προτάσεις μας. Και κάποια στιγμή μας ξαναφέρνετε πίσω τις προτάσεις και θέλετε να υπογράψουμε τελευταία στιγμή, χωρίς να διαβάσουμε καν τι έχετε φτιάξει. Οπότε Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Εμείς δεν λέμε ναι και το Συμβούλιο τα στυλώνει επί χρόνια. Αυτό είναι αδύνατον. Θέλουμε ισότιμη μεταχείριση με το άλλο νομοθετικό όργανο, το Συμβούλιο. Θα ήθελα και ένα κατάλογο, αν και θα... είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ μεγάλος με τα κολλημένα μέτρα. Λοιπόν, να ασκήσετε πίεση και στο Συμβούλιο. Και έρχομαι στο θέμα της εφαρμογής, αυτό το οποίο και όλοι οι άλλοι, γιατί νομοθετούμε, νομοθετούμε, νομοθετούμε και τα κρατημέλη εν τέλει δεν κάνουν τίποτα. Δακτυλικά αποτυπώματα, διαβατήρια, τα είπε και ο συνάδελφο Λέναρτ. Δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια έχουν περάσει από την εκπνοή τη προθεσμία. Δέκα χρόνια. Και τα μισά κρατημέλη δεν έχουν κάνει τίποτα. Η οδηγία για, τα, για την κακοποίηση παιδιών. 23 κράτη-μέλη δεν έχουν υλοποιήσει. Με συγχωρείτε. Ήρθε η Κομισιόν εδώ και μας πίεζε να το, να το περάσουμε γρήγορα και πού βρισκόμαστε. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Σλοβενία, Ισπανία, Γερμανία δεν έχουν εφαρμόσει. Λοιπόν, περισσότερη εφαρμογή. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Για το PNR. Δεδομένα ταξιδίου. Το δικαστήριο είπε ότι ο κανονισμό τότε δεν ήταν συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η συμφωνία με τι ΗΠΑ είναι ακόμα πιο μακριά από το ευρωπαϊκό δίκαιο, από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και δύο χρόνια μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει, δεν έχει προβεί σε νομική εκτίμηση, νομική αξιολόγηση. Γιατί? Και τέλος, αφού μιλάμε για πολιτικές ασφαλείας, θα ήθελα πραγματικά να μου πείτε μια συγκεκριμένη μορφή εγκλήματος με 2.500 θύματα το χρόνο, η οικιακή βία, η βία στο σπίτι, γιατί δεν αντιμετωπίζετε, γιατί δεν θεωρείτε θέμα δημόσιας ασφάλειας. Θα την συμπεριλάβετε στη, σας, στη γενικότερη σας στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σχινάλη, ο κύριος Φέστ, αναφέρατε την Ισλαμική τρομοκρατία. Υπάρχει μελέτη από τον Γαλλοκοινωνιολόγο Μπερνά Ρόζιε ο οποίος μας μιλάει ε, για μια εκστρατεία κατάληψης ουσιαστικά από τους ε, τρομοκράτες. Μας λέει ότι 150 πόλεις στη Γαλλία και μόνο είναι υπό τον έλεγχο των Ισλαμιστών και λέει ότι ανησυχεί και ότι είναι σαν να υπάρχει μια άτυπη συμφωνία, ένα σύμφωνο μεταξύ αριστεριστικών. Ε, εστερών οργανώσεων, κομμάτων και Ισλαμιστικών ομάδων. Και δίνει κάποια παραδείγματα που αφορούν τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, ίσως και την Ολλανδία. Το ερώτημά μου είναι τι μπορείτε να κάνετε για αυτήν την πέμπτη φάλαγγα των Ισλαμιστών που φοβούμαι υπάρχει μέχρι και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά η σχέση προσφύγων με έγκλημα, κυρίως σεξουαλικά εγκλήματα. Οι στατιστικέ είναι πολύ συγκεκριμένε στην Γερμανία, ξέρετε. Είναι ένα σκάνδαλο. Υπάρχει φόβο για καταγγελίε από τις ε, γυναίκες. Και τι γίνεται με του αριστερού που υποστηρίζουν του Ισλαμιστέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ φοβούμαι ότι πρόκειται για απειλή κατά τη ελεύθερη κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ, και Φέστ. Η πράσινη τώρα, η κυρία Τρεκ. Διαδικαστικό θέλετε να θέσετε. Είναι διαδικαστικά. Εδώ συμβαίνει κάτι το παράλογο. Πολλά πράγματα τα βάζουμε μέσα στην ίδια χωάνη. Ε, ε, πρόκειται για ένα λόγο μίσους κατά των αριστερών κομμάτων. Γίνεται και υπάρχει μία σύγχυση ως προς τα πάντα από τα κόμματα της δεξιάς. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για κάτι τέτοιο. Κυρία Έρνστ, θα λάβετε το λόγο σε λίγα λεπτά. Όταν λήξει ο γύρος των συντονιστών θα μπορέσετε να έχετε το λόγο. Να λάβετε το λόγο και να πείτε αυτά που θέλετε. Οι πράσινοι έχουν το λόγο, είναι η επόμενη εβδομάδα. Έχετε το λόγο, κυρία Ιντβέλτ είναι θέμα διαδικαστικό. Θα ήθελα να αποκρούσω τη σύνδεση που γίνεται μεταξύ άκρας δεξιάς και μετανάστευσης και κατάστασης των γυναικών. Όποιος και να προέρχεται από όποια θρησκεία παρενοχλεί τις γυναίκες. Είναι ένα θέμα δύο φύλων που αφορά τα δύο φύλλα δεν έχει σχέση με τις θρησκείες. Μπορούμε να μιλάμε για μουσουλμάνους, μπορούμε να έχουμε και ανθρώπους της άκρας δεξιάς οι οποίοι παρενοχλούν γυναίκες. Μην μου λέτε μένα τέτοια πράγματα. Εμείς, ε, ε, εγώ αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι είμαι γυναίκα και δεν μπορείτε να μου λέτε τέτοια πράγματα. Ωραία, εντάξει, εντάξει, αυτό το δέχεται η πλειοψηφία του σώματος, αλλά πρέπει να ακούμε τα μέλη, ό,τι και να λένε. Πρέπει να ακολουθούμε τον κανονισμό, αλλά όπως σας είπα, ας ακούσουμε τον, από τους πρασίνους. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι βλέπουμε την ανάγκη να μην προωθούμε ψευδοσυζητήσεις, να δούμε τα στατιστικά στοιχεία. Η Europol μας προβάλλει ακριβώς τα αντίθετα αυτά που λέει η άκρα δεξιά. Τώρα, θα θίξω τα ζητήματα που είχα σκοπό να θίξω ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κατά την ακρόασή σας είχατε πει ότι θέλετε να εισαγάγετε και τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα από την αρχή της εργασίας σας και όχι μόνο κατά την εφαρμογή. Πώς θα θέσετε σε εφαρμογή αυτή την προσέγγιση με βάση και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την παρακράτηση δεδομένων. Θα θέλαμε να μάθουμε τη δική σας προσέγγιση ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ως προς τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, ξέρετε ότι απασχολούν το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν το απασχολούν τόσο όσο άλλα εγκλήματα. Γι' αυτό γίνεται και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό απειλεί βεβαίως και τις επερχόμενες γενές αλλά και το περιβάλλον. Ποια είναι η στρατηγική της Επιτροπής επί του θέματος και πώς μπορείτε να ενσωματώσετε αυτή την στρατηγική ως προς ε, και το καθεστώς ε, της Europol, ως προς τον επαναπατρισμό των μαχητών. Ποια είναι η άποψή σας για την κατάσταση και την απειλή προς την ασφάλεια, ιδιαίτερα όταν χάνονται τα ίχνη τους στις χώρες που βρίσκονται. Δεν θα πρέπει να κριθούν στην Ευρώπη, να δικαστούν στην Ευρώπη και να ελέγχονται από τις δικαστικές υπηρεσίες. Από το ECR, ο κύριος Βάιμερς. Ναι, έχετε δίκιο, πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σχοινά, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας καταρχήν. Είπατε ότι ένας από τους τομείς προτεραιότητας είναι και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο ε, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να έχουμε την κοινωνική συνοχή που επιθυμούμε υπάρχουν ε, οι αδελφοί μουσουλμάνοι, μια οργάνωση που είναι κατά της ανεξίθρησκείας και σχετίζεται με την τρομοκρατία. Κατά την προηγούμενη θητεία είπαμε ότι δεν θα χρηματοδοτήσουμε καμία οργάνωση που έχει σχέσεις με την αδελφότητα των μουσουλμάνων. Και επειδή έχει σημασία η κοινωνική συνοχή. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε ομάδες που, είναι, που τάσσονται υπέρ του διαχωρισμού και του διχασμού. Ως Επίτροπος υπέρ του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής ε, δέχεστε ότι θα χρηματοδοτήσουμε ομάδες που τάσσονται υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών και ε, η χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να δοθεί προς οργανώσεις που υποσκάπτουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Η, κυρία Έρνστε έχει τώρα το λόγο από τη Γκουε και μπορεί να εκφράσει την άποψή μπορείτε να εκφράσετε την άποψή σας ελεύθερα. Δύο σημεία θα ήθελα να θίξω. Καταρχήν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια η οποία θα εκδοθεί τον Ιούλιο. Πολύ καλά είναι όλα αυτά, αλλά είχαμε πολλές στρατηγικές με το ίδιο όνομα τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η αξιολόγησή σας ως προς μέτρα ασφαλείας και ποια μέτρα μπορείτε να ε, απαλείψετε πριν φτάσετε σε νέα ε, θα το κάνετε αυτό ή θα έχετε ένα άλλο, ε, μία άλλη σωρία ε, μέτρων που θα προβάλλετε. Ως προς το PNR, τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να δράσει άμεσα η Επιτροπή. Πότε μπορούμε να έχουμε στοιχεία από εσάς ως προς τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μίλησε για τρομοκρατικές απειλές, για ε, ενδεχομένως επικείμενες ε, απειλές από την άκρα δεξιά. Είχαμε πολλά τέτοια επεισόδια στην Γερμανία με έναν φόνο που πολύ καλά γνωρίζετε και με συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι επικείμενοι κίνδυνοι από την άκρα δεξιά. Και αυτό το βλέπουμε και στις αστυνομικές δυνάμεις και στον στρατό. Θεωρείται ότι ελοχεύουν κίνδυνοι από την άκρα δεξιά και μέσα στον κρατικό μηχανισμό αλλά και εκτός αυτού. Υπάρχει κάποια στρατηγική σκέψη για την αντιμετώπιση της άκρας δεξιάς μέσα στα πλαίσια του κρατισμού και του κρατικού μηχανισμού, γιατί αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο της Γερμανίας. Ωραία λοιπόν. Έχω σημειώσει και τους υπόλοιπους που ζητούν το λόγο. Μπορώ να σας δώσω το λόγο σε όλους σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό μπορείτε. Ο κύριος Βίντσετ είναι ο πρώτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Σχοινά. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Μιλήσατε για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας. Προτείνω λοιπόν να μπούμε σε ε, λεπτομέρειες. Ε, συνεργασία στο χώρο της ασφάλειας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σχέδιο εντολής Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε τρία σκέλη. Το πρώτο πακέτο που είναι γενικές διευθετήσεις, το δεύτερο είναι οικονομικές και το τρίτο είναι της ασφάλειας. Και αυτό βέβαια είναι και το θέμα που απασχολεί την ΛΥΜΠΕ. Γιατί έχουμε τις κυβερνοεπιθέσεις, την παραπληροφόρηση, το οργανωμένο έγκλημα, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Εσείς πώς βλέπετε να συνδέονται ίδια πραγματεύσει τα οικονομικά θέματα με το Ηνωμένο Βασίλειο και πόσο στεναρά θα σταθούμε έτσι ώστε η συνεργασία στα θέματα της ασφάλειας θα είναι κομμάτι του πακέτου και εκεί θα αντιπροσωπεύονται και τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Εκτός μικροφώνου Επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε 10 λεπτά πρέπει να φύγω, οπότε φοβάμαι πως θα φανώ αγενής, γιατί θα φύγω πριν απαντήσετε, αλλά να μιλήσω πρώτα για τα 5G. Να σας πω πως κάνατε μια αξιολόγηση εξαιρετική. Τι θα γίνει μετά τι θα γίνει σε επίπεδο κρατών μελών και στι αποφάσει που θα λαμβάνουν για την εφαρμογή του 5G. Κάποιοι έχουν προχωρήσει περισσότερο. Κάποιοι έχουν επιτρέψει ήδη εταιρείε να συμμετέχουν σε αυτή τη τεχνολογία. Πιστεύετε πως υπάρχουν ασφαλή τμήματα ε, στο 5G. Γιατί όλοι πρέπει να είναι διασυνδεδεμένοι. Μήπως δεν πρέπει να επιτρέψουμε κανένα κίνδυνο να εισέλθει. Και όλοι μιλάνε για την ανακοίνωση για την τεχνητή νοημοσύνη. Πέραν των ηθικών κανόνων, πιστεύετε πως θα πρέπει να ποινικοποιήσουμε κιόλα. Γιατί είναι τεχνολογία η οποία στα ε, λάθος χέρια μπορεί να κάνει πολύ κακό. Και τελευταία ερώτηση, Europol. Εσείς θεωρείται στην ε, μεταρρύθμιση της Europol να έχουμε και ένα δικαίωμα πρωτοβουλίας της Europol να στρέφεται προς τα κράτη-μέλη και να θέλει, θέλουν να συμμετάσχουν στις έρευνες. Ε, σκεφτόμουν την περίπτωση της Μάλτας και της μεγάλης συμβολής της Europol. Θα έχουν λοιπόν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν ε, άμεσα να επεμβαίνουν. Κυρία Γιοντσέβα, παρακαλώ, σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Είναι πολύ απογοητευτικό που λείπει κάτι. Η διαφθορά. Να σας υπενθυμίσω, πριν από 5 χρο... 10 χρόνια, ε, στο πρόγραμμα του Στοκχόλμης είχαμε τη μάχη κατά της ε, διαφθοράς και μετά εξαφανίστηκε από την ημέρησα διάταξη για την ασφάλεια. Και από ό,τι ξέρω και από τη νέα εσωτερική, ε, στρατηγική εσωτερική ασφάλεια δεν θα εμφανίζεται. Διαφάνεια λοιπόν μόνο στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Είναι καλό αυτό, αλλά όχι αρκετό. Η διαφθορά έχει και ένα κομμάτι που αφορά τις διοκτικές αρχές. Και είναι φοβερής η επιπτώση που έχει για κάποια κράτη στη δικαιοσύνη, στο, στην οικονομία. Και στη Βουλγαρία, σύμφωνα με την έκθεση της ε, σχετικής, ε, του σχετικού κέντρου, χάνονται 11 δις λόγω διαφθοράς τεράστιο ποσό το οποίο ε, χάνεται και σε διασυνοριακό έγκλημα. Θα δώσετε προτεραιότητα στο θέμα της διαφθοράς στα πλαίσια της στρατηγικής για την εσωτερική ασφάλεια και τα σκάνδαλα που σχετίζονται με τη διαφθορά έχουν αρχίσει και ε, πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Θα κάνετε κάτι. Γιατί μπορεί τελικά η διαφθορά να μετατραπεί στο νέο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής έτσι όπως πάμε. Τι θα κάνετε για να το αποφύγουμε και για να χειραφετήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα. Θα σας ακούσω online όταν απαντήσετε γιατί δυστυχώς και εγώ πρέπει να αποχωρήσω. Ο κύριος Μπράιορ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Εάν οι δημόσιες αρχές θέλουν να ψάξουν παράνομο περιεχόμενο, δεν έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ. Είναι διεθνείς ιδιωτικές εταιρείες με τους ε, αδιαφανείς ε, αλγόριθμους ή με τους ε, κλικά με, τους υπαλλήλους τους που, που εκπέμπουν κλικ είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να δεχτώ. Επίσης, η διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Τόσα χρόνια μετά από την απόφαση του ΔΕΚ, τι θα κάνετε, θα ξεκινήσετε διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν έχουν καταργήσει ακόμα τους νόμους για την αδιάκριτη, δια, τη χωρίς διακρίσεις, διατήρηση των τηλεπικοινωνιών δεδομένων. Τέλος, η αίσθηση της ασφάλειας είναι κομμάτι της στρατηγικής σας. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και σε περιπτώσεις που ο κόσμος αισθάνεται ανασφαλής βασιζόμενος σε μια εσφαλμένη εντύπωση του κινδύνου αγνοώντας ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ασφαλής. Θα το αντιμετωπίσετε. Ο κύριος Μπουσατέ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ισπανικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Επίτροπε που είστε εδώ. Καλό θα ήταν δεδομένη τη συζήτηση και των όσων έχουμε πει. Να σας πω πως για την προστασία του ευρωπαϊκού τρύπου ζωής να δώσει ένα σημειωματάκι ε, ε στους ευρωβουλευτές εδώ ε, γιατί πρέπει να σέβονται τον πλουρανισμό. Κάποιοι μιλάνε και τους φωνάζουν και κάποιοι άλλοι μιλάνε και τους ακούνε όλοι. Λοιπόν, Έχω δύο θέματα. Μιλήσατε σήμερα και εγώ είμαι πολύ υπέρ του να ε, μην επιτρέπουμε τη ριζοσπαστικοποίηση online και τον περιορισμό ε, του τρομακρατικού περιεχομένου online. Τι θα κάνετε για να ελέγξετε κάποιους ναούς στους οποίους ακούγονται οι πιο ακραίες εκφράσεις ε, για το σαλαφισμό, για τον τζιχαντισμό, για το βασαμπισμό. Τι θα κάνετε. Εκεί ριζοσπαστικοποιούνται οι πολίτες στην Ευρώπη, όχι μόνο στο ίντερνετ. Και για τις καταπατήσεις και τις κακοποιήσεις σεξουαλικές στην ε, Ισπανία ε, δυστυχώς έχουν κακοποιηθεί ε, ανήλικοι σεξουαλικά σε κρετικά ιδρύματα στις Βαλαιαρίδες νήσους. Τι θα κάνετε έτσι ώστε η ελευθερία των παιδιών να μην είναι μόνο θύμα του ίντερνετ αλλά και της πραγματικότητας των ε, αρχών κυδαιμονίας που κάθε άλλο παρά προστατεύουν τα παιδιά. Κύριε Ντέλη, Επιτροπέ, λίγο περισσότερο μπορείτε να μας πείτε πώς θα βελτιώσετε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Γιατί ακούμε για απειλές και ότι δεν αρκεί μια κεντρική προσέγγιση. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Μερικά τα πιο σημαντικά εγκλήματα, διασυνοριακά εγκλήματα των τελευταίων ετών, συνέβησαν γιατί δεν πήραμε αρκετά μέτρα. Οι αστυνομίε δεν ε, πήραν αρκετά μέτρα γιατί το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιούσαν οι αστυνομίε είχε παραθυράκια, τα λογισμικά δεν συνεργάζονταν μεταξύ του κλπ. Τι θα κάνει λοιπόν η Κομισιόν για να αντιμετωπίσει λίγο πιο σοβαρά το θέμα του διασυνοριακού εγκλήματο για το οποίο δεν κάνουν τίποτα οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Μετά, έχουμε εμπειρογνώμονε, ειδικού, επιστήμονε, οι οποίοι εντοπίζουν κάθε τόσο κενά παραθυράκια στα συστήματά μας και δυστυχώς φοβούνται, όταν, φοβούνται να, μιλήσουν ότι υπάρχουν αυτά τα κενά ασφαλείας. Θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Και για το 5G, κρίσιμο θέμα, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, Τι θα γίνει με την κρυπτογράφηση της μεταφοράς δεδομένων από συσκευή σε συσκευή. Αυτά είναι κρίσιμα θέματα. Θέλει η Κομισιόν κάτι να κάνει. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη γραμμή άμυνα για μα. Και ο ε, Γιώχανσεν είπε ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να προστατεύσουμε την παράνομη υποκλοπή δεδομένων στο 5G. Δεν θέλουμε κυρκόπορτες. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε περισσότερα για το πώς θα λειτουργήσει το πράγμα στην πράξη. Ο κύριος Ρουμπέρτη. Κύριε Αντιπρόεδρε, μιλώντας για οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία που συνδέονται, δεν θα πρέπει να μιλήσουμε και για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Έχουν μεγάλη σημασία και δεν αναφερθήκατε σε αυτές τις πτυχές. Η ίδια η Επιτροπή πέρσι συνέταξε μία έκθεση μιλώντας για ανεπάρκειες σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνετε για να βελτιώσετε την κατάσταση σε πολλές χώρες ως προς αυτή την ανακύκλωση και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας γιατί και οι σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεγάλη σημασία κατά αυτής της ε, ανακύκλωσης, γιατί γίνεται λόγος για την ε, δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας με ανταλλαγή απόψεων. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, Φέτος η Eurojust γνώρισε μία μεγάλη μείωση κονδυλίων για τις δραστηριότητές της. Σας φαίνεται αυτή η δραστική μείωση της χρηματοδότησης της Eurojust συμβατή με την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ο κύριος Σασμάνη. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ, Πρόεδρε, που ήρθατε. Να ρωτήσω και εγώ κάτι που μας ανησυχεί. Εδώ και πολλά χρόνια στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο έχουμε μια συζήτηση για τις ε, παρεμβάσεις από τρίτες χώρες, ε, οργανώσεις, ε, θεσμούς στην κοινωνία μας που θέλουμε να σταματήσουμε. Κάποιες χώρες παρισφρίουν σε αυτές τις οργανώσεις, στέλνουν ρίζος παστικοποιημένα άτομα, δρομολογούν αυτό που ονομάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτά αποσταθεροποιούν την κοινωνία μας, καθώς και την ανεκτικότητα και την... το χαρακτήρα της κοινωνίας μας, που είναι μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Τι θα κάνουμε με αυτά τα μέτρα κατά των αποσυστικών τάσεων κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ θα παίξει κάποιο ρόλο. Και ε, συγκεκριμένα εσείς θα θέλετε να κάνετε κάτι στον τομέα. Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στα τρικά γεγονότα του Christchurch στην Οκένια, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στους αντίποδες, όπως λέμε. Αλλά θυμάστε και τι έγινε στο Ζάμεντεμ και στο Μάλμπεκ, μερικά χιλιόμετρα και μερικές εκατοντάδες μετρά μακριά, αντίστοιχα. Θυμηθείτε το Στρασβούργο, πώς βρήκαν εκεί το θάνατο κλπ. κλπ. Υπάρχει ένας ιστοτοπός religionforpeace.com Διαβάζουμε εκεί για τις σχετικές επιθέσεις τα θύματα στην Ευρώπη. Αλλά γιατί να πάμε πραγματικά στην Νέα Ζηλανδία. Ε, δείτε τις επίσημες στατιστικές των Σουηδικών, για παράδειγμα, αρχών. Η Σουηδική Ραδιοφωνία τα έχει δώσει αυτά. Δίνει επίσης ε, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 58% των δραστών δεν είναι Ευρωπαίοι. Αυτά τα λέει η δημόσια σουηδική τηλεόραση. Μετά μου λένε ότι εγώ διασπείρω ψευδοειδήσει. Αλλά δεν ξέρω, θα κατηγορήσετε τους Σουηδού, στη Σουηδική Ραδιοφωνία ότι ε, λέει ψέματα. Λοιπόν, θα μιλήσω γερμανικά, λέει η κυρία Βόλαθ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Frontex. Εδώ έχει να κάνει πολλή δουλειά. Είναι ο οργανισμός ο οποίος δραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο βάσει των στοιχείων του κ. Μισελ, του Πρόεδρου του Συμβουλίου. Τα κονδύλια δυστυχώ για τον Frontex θα μειωθούν κατά περίπου 40%. Είναι ακριβής αυτή η πληροφορία. Πιστεύω ότι ε, βάλετε αυτήν την ε, στιγμή. Πιστεύω ότι αν χρηματοδοτηθεί σωστά θα είναι μία από τις λύσεις για την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, όπου γνωρίζουμε ότι έχουμε προβλήματα, έχουμε αποθήσεις, έχουμε ε, βίαιη συμπεριφορά, δυσκολία πρόσβασης στις διαδικασίες, βολής ασύλου κλπ. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση αυτή και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου προκειμένου στα σύνορα. Ευχαριστώ. Και εδώ. Όχι, δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Νομίζω μιλήσατε. Όλοι έκλεισε ο κατάλογος. Ποιος άλλος είναι. Κύριος Παπαδάκης. Γρήγορα παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, κύριε Σκηνά, Στη συζήτηση διαφάνηκε πώς αξιοποιεί η ακροδεξιά ε, όλη αυτή την πολιτική καταστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα σύνορα, γιατί ακριβώς ε, πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θεωρεί ε, ότι εμπλέκεται στην ασφάλεια σύνορων οι, προ, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Γιατί διαμορφώνεται η αναβάθμιση του Frontex με 10.000 στα σύνορα στην Ελλάδα, διαμορφώνεται κατάσταση ε, απαράδεκτη με τα λεγόμενα πλωτά φράγματα που ε, στείνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα ελληνικά νησιά και τα κλειστά κέντρα. Μια πολιτική άγριας καταστολής που συνοδεύεται ταυτόχρονα με αναβάθμιση της παλιότερης αποστολής Σοφία στη Λιβύη που διαμορφώνει ένα εκρηκτικό έδαφος που στοχεύει απέναντι στην καταστολή των μεταναστών και των προσφύγων, θύματα των πολέμων που υλοποίησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί της. Άρα απέναντι σε αυτή την πολιτική ε, που εγκλωβίζει στα ελληνικά νησιά ε, με τον κανονισμό του Δουβλίνου και με την απράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έχει τεράστιες ευθύνες και οι ελληνικές κυβερνήσεις και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς τοποθετήσετε λοιπόν απέναντι στην ένταση της καταστολής απέναντι στους πρόσφυγες και μετανάστες. Πιστεύω ότι μιλήσαμε όλοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Σινά εκ των προτέρων, ο οποίος σημείωσε όλες τις ερωτήσεις. Σας υπενθυμίζω όμως ότι έχουμε κι άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη, το οποίο είναι και ιδιαίτερος τεχνικό. Έχουμε μια τελευταία ζήτηση λοιπόν επί 45 λεπτά. Λοιπόν, 15 λεπτά για το θέμα αυτό. Να κλείσουμε παρακαλώ. Δεν θα είναι εύκολο. Ευχαριστώ και τον προτέρων. Κύριε Σχοινά, να ευχαριστήσω πρώτον εσάς που προφέρετε σωστά το όνομά μου. Είστε ένας από τους λίγους, για να μην πω μοναδικός που είπε Σχοινάς. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Με την επιχείρηση Σοφία. Δυσκολεύομαι να σχολιάσω την χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Πολύ μάλλον διότι η Σοφία Β δεν, ξέρω πώς θα ονομάζεται αυτή η επιχείρηση. Θα είναι μια επιχείρηση ΚΕΠΑ. Εκτός δηλαδή των αρμοδιορίτων της κοινότητας. Πιστεύω ότι έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσους άλλους συμμετέχουν για να επιτηρούν το εμπάργκο ώστε να εφαρμοστούν τα συμπεράσματα της διάσκεψης του Βερολίνου στην οποία συμμετείχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χρόνος πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχει η επιχείρηση στις, στα ρεύματα μεταναστών και είμαστε έτοιμοι να εκτιμήσουμε αυτές τις επιπτώσεις, επιπτώσεις επί της μετανάστευσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών νομίζω είναι αρκετά σοφοί. Γνωρίζουν ότι πρόκειται για κάτι δύσκολο. Και φυσικά πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο δεν θα πετύχει τα πάντα εν μία νυχτή. Λοιπόν, για την λειτουργική συμβατότητα που είναι σημαντική για εσά και πολύ σωστά. Το είπα εξ αρχής ότι θα υποστηρίξουμε την ε, λειτουργική συμβατότητα, την διαλειτουργικότητα, όπως λέμε, με κονδύλια, με συνεχείς αξιολογήσεις, εκθέσεις και από εκεί πέρα θα δρομολογήσουμε τις διδικασίες υπεραβάση, αν χρειαστεί. μίλησε με τον διευθυντή ε, Γιουλίση, μάλιστα, ο οποίος με διαβεβαίωση για την ε, βολησή του, τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί αμέσως. Για τα βιομετρικά στοιχεία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η πρόταση της Eurodac είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως γνωρίζετε. Θα τη συζητήσουμε. Είμαι βέβαιος ότι θα πάμε παρακάτω. Ε, και συμφωνώ με τους περισσότερους από εσάς ότι χρειαζόμαστε συστηματικές καταγραφές. Για το 5G Ήμουν ε, στο Μόναχο το Σαββατοκύριακο στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου και ξεπλάγει θετικό βλέποντας ότι η προσέγγιση μας δέκα μέρες πριν της δέσμης μέτρων της Ιρελιοθήκης έγινε αποδεκτή ως ένας πραγματικά ευρωπαϊκός τρόπος αντιμετώπισης όλων των σχετικών ζητημάτων. Έχουμε πολλά διαφορετικά ζητήματα, τα οποία απτώνται της ασφαλείας, αλλά έχουμε και σοβαρές γεωπολιτικές επιπτώσεις όσον αφορά τους παρόχους των λύσεων του συστήματος που παρουσιάσαμε, μιας αρχιτεκτονικής αν θέλετε, η οποία ξεκινάει από την εργαλειοθήκη αλλά προβλέπει και άλλα με τα επόμενα βήματα που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, να παρακολουθεί τους κινδύνους. Τα κρατη έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν κινδύνους για κρίσιμες υποδομές. Κύριε για την ανάγκη και την υποχρέωση εφαρμογή υλοποίηση αυτών που υποσχόμαστε. Μα κοιτάξτε, ε, εγώ θα είμαι βασιλικό τώρα του βασιλέο ε, διότι είπα, θα είμαστε αμήλικτοι. Θα είμαστε αμήλικτοι. Είμαι ταγμένο ε, με τρόπο αδύρυτο στην εφαρμογή, στην υλοποίηση, στην πράξη αυτών που αποφασίζουμε. δεν θα συνεχίσουμε να αερολογούμε χωρίς να εφαρμόζουμε. Επίσης για την ε, μελέτη υλοποίησης είναι υπό εξέλιξη, θα το ξαναδούμε. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει λόγος να το ξαναδούμε, να πάμε παρακάτω πέρα από την ε, μελέτη αυτή, θα προχωρήσουμε. Για την των παιδιών, σεξουαλική εκμετάλλευση κλπ. Υπάρχει εντολή. Πήγα στη Europol πρόσφατα μάλιστα και συζήτησα, νομίζω ότι έχουν πολλές επιτυχίες στον τομέα αυτών. Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε. Μπορούν να συνεργαστούν με ιδιωτικές εταιρείε και φυσικά προκειμένου πρέπει η κοινωνία των πολιτών, οι επιχειρήσει, ε, τα σώματα ασφαλεία και άλλοι φορεί, υπάρχει τεχνολογία κλπ. Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα. Για την ριζοσπαστικοποίηση, το δίκτυο RAN βεβαίως συνεχίζει να είναι στο κέντρο της δράσης μας. Εκεί συνεργάζονται οι ειδικοί. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, έχουμε δώσει 60 εκατομμύρια στο έργο αυτό. Όμως στη Μεσαφής δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Δεν λύνουμε το πρόβλημα πατώντας ένα κουμπί από τις Βρυξέλλες, έτσι για να εξαφανιστεί για να εξαφανιστούν τα ριζοσπαστικά στοιχεία. Χρειάζεται δουλειά σε όλα τα επίπεδα, Ξεκινώντα από τις φυλακέ, τα σχολεία, τι ε, τοπικές κοινωνίες, ε, το περιφερειακό επίπεδο, τις εκκλησίες. Πολλή δουλειά με όλους που μπορούν να βοηθήσουν. Για την ερώτηση τη κυρίας Ιντβέλτ. Έκανε, έγιναν ορισμένες αξιόλογες υποδείξεις για το σχήμα one-in, one-in. Συμφωνώ αν βρείτε ένα τρόπο να ενταχθεί στα συμπεράσματα του Σύμβουλου Υπουργών, έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί διαφορετικά, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα νομίζω ευρηματική σε θέματα δικής μου ειδικότητα. Για το PNR γίνονται προετοιμασίες, ξέρουμε πόσο λεπτό είναι το θέμα. Θα γίνει και μία νομική ανάλυση που θα υποβληθεί τους επόμενους μήνες. Είναι δέσμευση και καλύτερα να γίνει νωρίτερα παρά αργότερα. Δεν θα απαντήσω στον κύριο Φέστ, δεν είναι σκόπιμο. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι ήμουνα στο Auschwitz για την επέτειο των 75 ετών της απελευθέρωσής του, δηλαδή με τους επικεφαλείς επικεφαλείς κρατών και είπα ότι οι δαίμονες του παρελθόντος της ευρωπαϊκής ιστορίας δεν σχετίζονται με τους μετανάστες. Δεν υπήρχαν μετανάστες στο Auschwitz. Ως προς αυτά που είπε η κυρία Ρίκμον, ε, για την παρακράτηση δεδομένων. Η θέση μας είναι σαφής. Θα περιμένουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα γίνουν και μελέτες βιωσιμότητας και για την καλύτερη ρύθμιση νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια ε, ανάλυση αντικτύπου. Δεν προτείνουμε μέτρα παρά μόνον αν είμαστε σίγουροι ότι βασίζονται σε αδιάσυστα στοιχεία. Το ερώτημα του συναδέλφου από το ECR για, τον, ε, για τη συνδεσιμότητα μεταξύ ε, χρηματοδότησης και τρομοκρατικών στοιχείων. Ε, αντίθετα, εμείς έχουμε πολλαπλούς ελέγχους πριν από τη χρηματοδότηση και αν έχετε στοιχεία προς την αντίθετη κατεύθυνση θα ήθελα να τα μάθω. Πώς ε, επίσης αξιολογούμε την ασφάλεια στην Ευρώπη. Έχουμε 20 εκθέσεις προόδου που ε, δημοσιεύουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και ε, έχουμε κάνει και μία κατάδυση, θα μπορούσα να πω έτσι, ώστε να, συμμετάσχουν, να συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες της Επιτροπής για τη γενικότερη στρατηγική μας, η οποία θα συνοδευτεί από μελέτη αντικτύπου που θα δημοσιευτεί φέτος. Ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα ήθελα να μιλήσω για το Brexit. Νομίζω ότι είναι μέρος της αρνητικής μας ατζέντα. Εγώ θα προτιμούσα να μιλήσω για τη θετική μας ατζέντα, αλλά εφόσον με ρωτάτε, θα ήθελα να πω ότι η συνέχεια των διαπραγματεύσεων θα γίνει υπό την Task Force του Μισελ Μπαρνιέ που θα ε, γίνει ε, με τα κράτη-μέλη και με τις συναρμόδιες γενικές διευθύνσεις και θεωρώ ότι χρειάζεται μια εταιρική σχέση ασφαλείας για ότι ε, φυσικά δεν διακυβεύεται η ασφάλεια για, ε, για να υπηρετήσουμε οικονομικές σκοπιμότητες. Ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα και μετράω τα λόγια μου, αλλά μπορώ να πω ότι γράψαμε ιστορία στο Διευθυντήριο με αυτή τη διαδικασία ευρωπαϊκής πλαισίωσης για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Βεβαίως δεν είμαστε και η μόνη δύναμη ανά τον κόσμο που πράττει κάτι τέτοιο. Τα ζητήματα που θέτουμε, ποιος είναι ε, ο υπεύθυνος των αλγορίθμων και ε, πώς, κατά πόσο θα ξέρουμε ότι οι αλγόριθμοι δεν θα είναι στα ε, χέρια των εμπειρογνωμόνων, αλλά θα γνωστοποιούνται και ευρύτερα. Ξέρετε ότι οι απαντήσεις της ΣΥΠΑ, η απάντηση ΣΥΠΑ είναι φανερή και ε, η απάντηση βεβαίως είναι και η Κίνα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το στοιχείο, αυτό το ιστορικό ε, ε, βήμα από εμάς και θα ήθελα όλα τα δίκτυα να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης για να φτάσουμε σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Ως προς την εντολή της Europol θα πρέπει να μιλήσουμε για αναδιόμενες απειλές, συνεργασία με χώρες και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Ε, για την ερώτηση της κυρίας Γιόντσεβα για την διαφθόρα στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης και του εξαμήνου έχουμε ειδικέ συστάσεις του Συμβουλίου για και οκτώ κράτη-μέλη έχουν λάβει ειδικέ συστάσεις για τη διαφθορά, για το κράτος δικαίου και θα αναθεωρήσουμε και το ποινικό δίκαιο ως προς τη ριζοσπαστικοποίηση, το συζητήσαμε το θέμα, θα πρέπει να συνδράμουν και οι τοπικές αρχές, γιατί δεν είναι ένα θέμα που αφορά τις Βρυξέλλες, αποκλειστικά για την κρυπτογράφηση. Έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση διαπραγμάτευση και όπως σας είπα, οι πολίτες μας θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς ε, και να σεβόμαστε την ιδιωτικότητά τους. Ως προς το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, αύριο προβλέπεται ένα έκτακτο συμβούλιο. Υπάρχουν δύο σχολές, θα μπορούσα να πω. Πολλοί πιστεύουν ότι φτάνουμε σε αυτό το πολιετές και άλλοι που θεωρούν ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, εγώ στέκομαι σαν τον κολοσσό της Ρόδου ανάμεσα στις δύο σχολές. Ο Σαρλ Μισελ έχει προχωρήσει και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία συνένεση ως προς τα δικά μας θέματα. Επειδή τώρα δίνουμε τελική μορφή στο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου θα θέλαμε οι συνομιλητές μας να γνωρίζουν ότι οι φιλοδοξίες συνοδεύονται από δράσεις με μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη, με πόρους και σχέδια. Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ε, τομείς μετανάστευσης και ασφάλειας μέσα στα πλαίσια αυτής της ασυμμετρίας προσδοκιών και πραγματικότητας, γιατί κατ' εξακολούθηση μιλήσαμε για ευθύνη και βεβαίως για τα σύνορα και διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια Frontex με 10.000 συνοριοφύλακες και να δούμε ότι δεν μπορούμε να συνδράμουμε νομοθετικά. Η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν που θα εκπροσωπήσει αύριο την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γνωρίζει καλά τις ευαισθησίες που υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα. Ο οποίος όπως και στο παρελθόν ε, προσπαθεί να μου πει ότι το γεγονός ότι η ακροδεξιά ε, καπηλεύεται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Ε, εγώ αντιστρέφω αυτό το επιχείρημα και λέω ότι η ακροδεξιά περιμένει να δει αν τσιμπάμε εμείς σε αυτό που ε, πιστεύει, περιμένει να δει εμείς να ενοχλούμαστε για να θεωρήσει τον εαυτό της νικητή. Ε, δεν με εντυπωσιάζει κανένα από τα επιχειρήματα της ακροδεξιάς. Εγώ πιστεύω στη διαχείριση του μεταναστευτικού χρειαζόμαστε καθαρό μυαλό, ψυχραιμία, σύνεση, όχι κραυγές και κυρίως όχι ε, εύκολες λύσεις. Ζήσαμε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης ε, το φαινόμενο πολλών να προτείνουν απλές ή απλοϊκές λύσεις σε πολύ σύνθετα προβλήματα και απέδειξε η ιστορία ότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν άδικο. Οι καλές λύσεις είναι οι μεσαίες λύσεις, οι ουσιαστικές λύσεις, αυτές που παίρνουν υπόψη τους όλες τις πλευρές του προβλήματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε για αυτό το διάλογο για να δούμε την στρατηγική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβουμε ό,τι χρειαστεί υπόψη στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου σας. Όπως είπατε υπάρχουν περιθώρια συζήτησης. Κύριε Ρομπέρτη, δεν ε, μπορείτε να αντιδράσετε τώρα. Μα τι πιστεύετε για, την Ευρωπαϊ... τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό κατά της ανακύκλωσης και τη Eurojust. Το πρώτο τελευταίο που είπα είναι ότι στις διαπραγματεύσεις για τις ΠΔΠ θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε στόχους και φιλοδοξίες με κονδύλια και δράση. Αυτό καλύπτει και τούτη την υπηρεσία και ξέρετε πως ανήκει περισσότερο στα θέματα της ε, ε, Βέρα Γιούροβα και του κυρίου Ρέινχαρτς και όχι στα δικά μου. Επίσης, Συνάδελφοι, έχουμε ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ πολύ, δείξτε υπομονή, μείνετε στην αίθουσα, γιατί ακόμα έχουμε πολλά να πούμε για το σχέδιο έκθεση, για ένα πολύ τεχνικό θέμα, ε, το οποίο σίγουρα θα χρειαστεί να παρακολουθήσουμε για κάποια λεπτά, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα για να κλείσουμε και με τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Συνάδελφοι, μας πιέζει ο χρόνος. Έχουμε ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν να ε, καθίσετε και να μην μιλάτε. Καθίστε σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, μην μιλάτε στην αίθουσα. Έχουμε να κάνουμε με την απόφαση, την εφαρμοστική, για να ξεκινήσει η ανταλλαγή αυτοματοποιημένη δεδομένων για τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα με το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι μόνο δακτυλικά αποτυπώματα. Ξέρετε πως έχει κατάσταση το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γίνει σύντομα τρίτη χώρα για όλα τα θέματα. Θα συμβεί αυτό 31 Δεκεμβρίου, οπότε από τον Ιανουάριο θα είναι τρίτη χώρα, πιέζει ο χρόνος, γιατί χρειάζονται διαπραγματεύσεις, έχουμε 10 μήνες μπροστά μας για να συμφωνήσουμε για την ε, επόμενη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου και υπό αυτές τις συνθήκες, οι οποίες είναι εξαιρετικά πιεστικές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει μία εφαρμοστική απόφαση για την ανταλλαγή αυτοματοποιημένων δεδομένων και το σχέδιο αυτό ε, του Συμβουλίου για τέτοιου είδους δεδομένα, δηλαδή δαστηλοσκοπικά, ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μία ψηφοφορία συμβουλευτική. Να σας πω πως το Δεκέμβριο του 19 μας ζητήθηκε να καταθέσουμε μία γνώμη για το σχέδιο αυτής της πράξης και το συνομότερο όχι, ε, δηλαδή να περάσουμε το όριο των τριών μηνών. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ε, στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου. Άρα λοιπόν πρέπει να βιαστούμε να επιταχύνουμε. Θέλουμε εδώ λοιπόν να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την Προεδρία του Συμβουλίου για το πώς έχει αυτή η εφαρμοστική απόφαση ε, με την ανταλλαγή πληροφοριών, το σκεπτικό πάνω στην οποία βασίστηκε. Εγώ είμαι εισηγητή σας εδώ, είμαι ο εισηγητή σας. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως το Συμβούλιο στην πρότασή του φωτίζει το γεγονός πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν σκοπεύει να ε, συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της ε, απόφασης στην ΠΡΥΜ. Τα θυμόσαστε και θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση για το πώς θα χρησιμοποιεί ε, και θα συμπεριλαμβάνει δεδομένα για υπόπτους, γιατί έχουν πει δεν θα το κάνουν μόνο σε καταδικασμένα άτομα. Μόλις λοιπόν λήξει η μεταβατική περίοδος, δηλαδή η τέλη Δεκεμβρίου, το Ηνωμένο Βασιλείο αποτελεί πλέον πλήρως τρίτη χώρα και αυτό σημαίνει πως νομικά ομιλώντας χρειαζόμαστε να εγκρίνουμε ένα νέο νομικό εργαλείο. Έτσι κι αλλιώς. Αν εγκριθεί η εφαρμοστική απόφαση, δεν σημαίνει πως θα έχουμε ένα καθεστώς ε, θα έχουμε απλώς μία μεταβατική ε, ε, συμφωνία για το πώς μπορούμε να ανταλλάσσουμε δεδομένα με μία χώρα με την οποία τρέχουν και πιεστικές διαπραγματεύσεις χωρίς καμία εγγύηση πως θα έχουμε αμοιβαιότητα και πως θα συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κυρίως με αυτά τα οποία είχαμε στην δικασία της ΠΡΙΜ. Αυτά. Να, μας, να ακούσουμε λοιπόν την κυρία Πέτκοβιτς που είναι εκπρόσωπος κρατικής προεδρίας για να μας εξηγήσει το σκεπτικό για να δούμε και συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία έχω εγώ κατά νου. Θέλω λοιπόν σας παρακαλώ, επειδή είμαι εισηγητή και γι' αυτό χρησιμοποιώ τόσο χρόνο εδώ, θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω πως 12 Φεβρουαρίου Πρόσφατα δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια ενέκρινε ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε από 543 μέλη του Κοινοβουλίου. και τις μεγαλύτερες ε, κοινοβουλευτικές ομάδες εδώ. Και εκεί δηλώσαμε το εξής, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα της, ε, των βάσεων ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να συμμετέχει στις υπηρεσίες, στις υπηρεσίες και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Και χρειάζεται να τοποθετήσουμε τις ε, δικλείδες ασφαλείας με παρακολούθηση και ασφάλεια έτσι ώστε τα προσωπικά δεδομένα να την χάνουν αντίστοιχου υψηλού επίπεδου προστασίας από αυτά τα οποία προβλέπει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και δεν έχουμε λάβει τέτοιες εγγύησεις. Οι δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό κύριο Τζόνσον λένε πως έχει σκοπό να θέσει τα δικά του πρότυπα για τα δεδομένα τα οποία δεν θα αντιστοιχούν σε αυτά που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όχι. Έτσι το είπανε. Απερίφραστα. Οπότε αυτό που λέω είναι πως μας διακατέχουν ε, σοβαρές ανησυχίες πως δεν θα έχουμε αυτή την αμοιβαιότητα μέσα στο χρόνο που θα μας επιτρέψει να κάνουμε μια αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων γιατί τα πρότυπα αυτά δεν θα τα έχουμε ε, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που χρειαζόμαστε, το οποίο σημαίνει είναι απίθανο αυτά τα SAS, τα SIS συστήματα που είναι τα συστήματα ανταλλαγή, τα συστήματα πληροφοριών Schengen δεύτερης γενιάς, τα οποία καταπάτησε ε, ξεκάθαρα το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνοντας δεδομένα σε τρίτες χώρες, αυτά λοιπόν δεν θα ε, γίνονται σεβαστά και δεν θα ε, ε, βελτιωθούν αυτά τα σφάλματα τα οποία έχουμε διαπιστώσει εμείς πως υπάρχουν και τα ελλείμματα. Άρα λοιπόν και γι' αυτό έχουμε καταλήξει σε αυτή τη σύσταση που κάνω και θα ήθελα η εκπρόσωπος της Κροατικής Προεδρίας μας να μας πει τι θα γίνει με το θέμα του DNA και με την καταχώρηση των οχημάτων γιατί δεν βλέπω πουθενά να γίνεται κάτι αντίστοιχο με αυτά που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο Άρα λοιπόν έχουμε μία ακόμα πρόκληση και ένα ακόμα πρόβλημα για το πώς μπορούμε εμείς να εγκρίνουμε αυτή την εφαρμοστική απόφαση. Ας μιλήσει η Κροατική Προεδρία και μετά μπορούμε και να το συζητήσουμε. Κροατική Προεδρία σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Good everyone. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Εξ ονόματος της Προεδρίας θα ήθελα να σας παρουσιάσω την πρόταση του Συμβουλίου ως προς την πρόταση εφαρμοστικής απόφασης για την ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών στοιχείων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Συμβούλιο υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στις 12 Δεκεμβρίου 2019 το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης. Θέλω να τονίσω ότι η έγκριση είναι δυνατή από νομική και τεχνική άποψη και κυρίως, κυρίως από επιχειρησιακή άποψη, από την άποψη της εσωτερικής ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, μετά από την ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ανταλλαγή Δεδομένων εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περίοδου με την επιφύλαξη μετά της συμφωνία αποχώρησης και δι του άρθρου 127. Το Ηνωμένο Βασίλειο από την πλευρά του είναι έτοιμο να εφαρμόσει τη σχετική απόφαση. Το Συμβούλιο αξιολόγησε την εφαρμογή της Συμφωνίας για τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε θετικά Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο σύνταξε την εκτελεστική απόφαση η οποία εστάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους σκοπούς της διαβούλευσης. Μην ξεχνούμε τα εξή. Δεδομένη τη πρακτική και επιχειρησιακή σημασία τη συμπερίληψη των προφίλ υπόπτων στο πλαίσιο τη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων για του σκοπού τη δημόσια ασφάλιση και δι για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματο. το Συμβούλιο ζήτησε αναθεώρηση από τον Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την 1η Μαρτίου όσον αφορά την συμπερίληψη των προφίλ υπόπτων. Κάτι πολύ βασικό και το οποίο περιλαμβάνει την ανταλλαγή στοιχείων DNA. Όσον αφορά την ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων και άλλων, δεν ε, παρά την ε, ανάλυση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μας έχει ενημερώσει το τι θα κάνει. Το Συμβούλιο λοιπόν θα επανεκτιμήσει την κατάσταση με στόχο την συνέχιση ή διακοπή της ανταλλαγής δακτυλοσκοπικών δεδομένων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Συμβούλιο θα εκτιμούσε πολύ αν το, Ηνωμένο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκλεινε τη διαδικασία γρήγορα για να μπορέσει να προχωρήσει η έγκριση της σχετικής απόφασης, της εκτελεστικής δηλαδή απόφασης. Όσο αφορά τις ανταλλαγές DNA, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επιχειρησιακά έτοιμο από τα μέσα του Ιουνίου του 19. Πάνω από 50.000 αναζητήσεις έγιναν σε συνεργασία με 7 κρατημέλη τα οποία ήταν ήδη συνδεμένα από τα μέσα του 19. Τώρα, γιατί το Συμβούλιο θέλει να εκτελέσει, να υλοποιήσει μάλλον αυτή την εκτελεστική απόφαση για να ενισχύσει την εσωτερική ασφάλεια και να υποστηρίξει βεβαίω την εφαρμογή του νόμου. Η επιχειρησιακή εμπειρία με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην περίπτωση του DNA, έχει αποφέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πάνω από 50.000 διασταυρώσει παρήχθησαν κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2019. σε πάνω από 8.000 περιπτώσεις έγινε δυνατό να εντοπιστεί το άτομο βάσει του DNA του και μάλιστα πρόσωπα τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί προηγουμένως σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων. Παράδειγμα, σε 5.543 περιπτώσεις οι Γάλλοι από ίχνη που συνελέγησαν κατά τη διάρκεια ερευνών κατόρθωσαν να εντοπίσουν πρόσωπα τα οποία υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ίδιο στη Γερμανία. 3.763 μη εντοπισμένοι με αντίστοιχα γενετικά προφίλ βρέθηκαν και επιβεβαιώθηκε η ύπαρξή τους στα αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό δείχνει πόσο εξαιρετικά δουλεύει η βάση δεδομένων προύμ και πόσο ενισχύει την ιστορική ασφάλεια η ιστορική ασφάλεια στην Ένωση είναι υψής της σημασίας για όλους μας. Ακόμη και μία διασταύρωση, επιτυχημένη διασταύρωση προύμ με το Ερμένο Βασίλειο το 2020 θα συνέβαλε στην διελεύκανση σοβαρών εγκλημάτων ή εγκλημάτων αδικημάτων τρομοκρατίας στην περίπτωση βεβαίως ε, που υλοποιηθεί η απόφαση και συνεχιστεί η ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων. Τώρα, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιθυμούσε ενδεχομένω ε, να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην αλλάξει την νομοθεσία του. Θα ήταν, πιστεύω, στο, προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα χάσει το δικαίωμα να συμμετέχει στην ανταλλαγή δεδομένων που οι δείχνουν ότι θα υποφεληθούν όχι μόνο τα κρατημέλη, αλλά και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάνω από 3.300 μη αναγνωρισμένα προφίλ αντιστοιχίστηκαν σε βάσεις δεδομένων των κρατών μελών. Όσον αφορά τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν της μεταβατικής περίοδου, αυτές θα εξαρτηθούν από τις προσεχείς διαβουλεύσεις. Και για αυτό το θέμα δεν έχω παρά να δώσω τον λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σε σχέση με το θέμα όμως ε, της καταχώρησης σε ένα μητρό, θα ήθελα να ξέρω πώς έχει η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο επί του θέματος, διότι δεν φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει αυτό το πλαίσιο διασταυρώσεων DNA ε, πέρα από τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία όταν ζητηθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι ήδη απάντησα σε αυτή την ερώτηση. Θα σας δώσω και παραδείγματα. Σε σχέση με την ανταλλαγή δεδομένων DNA έχουμε 7 κράτη-μέλη που είναι συνδεδεμένα. 7, 7 κράτη-μέλη που είναι ο κύριος ε, Ρότσενμπεργκ που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έχει να μας πείτε σε σχέση με αυτή την ε, εκτελεστική απόφαση. Θα είμαι πολύ σύντομος ε, σε σχέση με την Επιτροπή. Λαμβάνουμε γνώση της έκθεσής σας και εμείς, όπως και εσείς, ε, πιστεύουμε στην απόλυτη αμοιβαιότητα ανταλλαγής στοιχείων με βάση τη σύμβαση ΠΡΟΥΜ, αλλά όπως φαίνεται είναι μία διαδικασία όπου επικεφαλής είναι το Συμβούλιο. Αν δούμε τώρα την απόφαση και σε σχέση με αυτά που είπε η Προεδρία μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι αποφάσεις πριν ισχύουν και κατά τη μεταβατική περίοδο που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα το Συμβούλιο στην εκτελεστική απόφαση θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ανταλλαγή αυτή προσωπικών δεδομένων δυνάμει της απόφασης ε, πρώην. Δεν πρόκειται για, ε, για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου και η αποτίμηση του Συμβουλίου είναι πολύ ακριβής και πιστική. Ως προς το μέλλον θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μετά το, το δημοψήφισμα του 2016 η Επιτροπή ε, ε, έχει μία προσέγγιση νομικού τύπου, όχι νομικιστικού, νομικού και εφαρμόζει τα δεδομένα με βάση ε, τους κανόνες που ε, θα ισχύσουν για το Ηνωμένο Βασίλειο για το υπόλοιπο του έτου και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση. Ως προς το ερώτημά σας για την ανταλλαγή στοιχείων DNA και την καταχώρηση οχημάτων, ε, έχουμε απόλυτα πιστικά στοιχεία ως προς τα δακτυλοσκοπικά στοιχεία δεν υπάρχει ανταλλαγή, γι' αυτό γίνεται και αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Και ως προς την καταγραφή οχημάτων δεν έχουμε ακόμα ανταλλαγή στοιχείων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί το σύστημα δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά κοιτάξτε, κατανοήσαμε την διαδικασία αυτή. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάθε δικαίωμα και καθήκον να αποστείλει ένα πολιτικό μήνυμα και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ε, αναλάβει αυτές τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε όταν το Ηνωμένο Βασίλειο μετατραπεί σε τρίτη χώρα θα πρέπει να συμμορφωθεί με αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Μία απόφαση θα πρέπει να ληφθεί. Το ζήτημα είναι να δούμε πώς έχει κατάσταση. Γιατί ναι, μιλάμε για ανταλλαγή δεδομένων. Αλλά από όσο ξέρουμε μόνο 7 κράτη-μέλη. Από τα 27 μόνο 7 κράτη λαμβάνουν ε, στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά με βάση την απόφαση πριν θα πρέπει εμείς να διαβιβάζουμε αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν υπάρχει αμοιβαιότητα με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, δηλαδή με τα υπόλοιπα 20 κράτη-μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της, γιατί είσαστε θεματοφύλακας της εφαρμογής του νομικού πλαισίου. Πώς θα έχει κατάσταση μετά τις 31 Δεκεμβρίου. από την 1η Πρώτου 21 το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μια τρίτη χώρα. Θα λαμβάνουμε στοιχεία, θα γίνεται ανταλλαγή. Ποια πίεση μπορούμε να ασκήσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο έτσι ώστε να προσαρμοστεί νομικά για να ανταποκριθεί σύμφωνα με τη ρήτρα αναθεώρησης που όρισε και εξήγησε το Συμβούλιο. Μιλάμε για την 15η Ιουνίου. Θα πρέπει να ανταλλάσσουν στοιχεία σε σχέση με υπόπτους. Έχουμε έξι μήνες, μιλάμε μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και μετά άλλους έξι για τη λήξη της μεταβατικής περίοδου. Τι θα, ποια θα είναι η πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτά τα δεδομένα και ποια στοιχεία θα ε, μεταβιβάζει. Μπορείτε να μας απαντήσετε. Λίγο εισηγητής, λίγο προεδρία, αλλά πριν πάμε στο δεύτερο γύρο, να ακούσουμε και τις άλλες ομάδες πώς βλέπουν το θέμα. Για να χωρίς μικρόφωνο ομιλητής. Έχουμε λίγα λεπτά. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα υπολοιπόμενα λεπτά. Λοιπόν, τι, τι θα γίνει, η ερώτησή μου είναι τι θα γίνει μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Ποιο θα είναι το νομικό καθεστώς και πώς θα φροντίσει η Κομισιόν να υλοποιηθεί, να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αφού φύγει εντελώς το Ηνωμένο Βασίλειο. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Εάν την πρώτη 2021 δεν υπάρχει νέα συμφωνία και έχει φυσικά εκπνεύσει η μεταβατική περίοδο, τότε σημαίνει ότι η σύνδεση με το σύστημα Πλουμ ε, πάβει. Μάλιστα. Σωστά. Οι σκιώδεις παρακαλώ. Κυρία Βαστιλίμα. Ευχαριστώ για όσα είπατε και να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Γιατί είχα ερωτήσεις που ήθελα να, να θέσω, αλλά ήδη απαντήθηκαν. Αν επιτρέπετε, Πρόεδρε, μια πολύ σύντομη εισαγωγή στα γαλλικά. στο συγκεκριμένο πλαίσιο να πω το εξή. Έχω θαυμασμό, μεγάλο θαυμασμό για το έργο του Μπαρνιέ. Πετύχαμε ενότητα ως 27. Γιατί το λέω αυτό. Διότι θεωρώ ότι οφείλουμε οι στάση μας να είναι αμέμπτη έναντι της Βρετανίας. πρέπει να σεβαστούμε τους Βρετανούς ως χώρα η οποία σε λίγο θα είναι τρίτη χώρα έναντι της οποίας όμως θέλουμε τις στενότερες δυνατές σχέσεις προς όφελος τόσο της Βρετανίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελα να διατυπώσω λοιπόν αυτή την σύντομη εισαγωγή στα γαλλικά και συνεχίζω στα αγγλικά. όσον αφορά το έγκλημα και την τρομοκρατία. Θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία να εξασφαλίσουμε καλή συνεργασία σήμερα ήδη από το, με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και μετά την εκπνοή της μεταβατικής περίοδου. Θέλουμε τον τόνο για την μελλοντική συνεργασία. Οφείλουμε να παραμείνουμε στενοί εταίροι προκειμένου περί της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν θα στέλνει αποτυπώματα από 9 εκατομμύρια καταδικασέντες πέραν των 5 εκατομμυρίων των οποίων το προφίλ DNA έχουν προκύψει από έρευνες. Όπως συμφωνήθηκε άλλωστε διαβοήθηκε το 2019. Η ανταλλαγή DNA με το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή αξιοποιείται και μάλιστα από περισσότερες χώρες από ό,τι νόμιζα ήξερα, τουλάχιστον Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, κατοχώρες, Αυστρία. Το θέμα είναι αυτή, ότι αυτή η ανταλλαγή είναι χρήσιμη και τους δύο. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει την μεγαλύτερη βάση δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάση DNA και ε, δακτυλοσκοπικών δεδομένων. Πιστεύω ότι εμείς θα βγαίναμε χαμένοι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μας επέτρεπε πλέον πρόσβαση δικά του δεδομένα. Πολύ περισσότερο από ότι θα βγαίνει χαμένο το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μ' αρέσει τώρα το χαμένο ή το ποιο τιμωρεί ποιον, αλλά έτσι έχει κατάσταση. Επίσης, είναι απολύτω αληθέ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε στην ομάδα Μπερνιέ πολύ σαφή διαπραγματευτική εντολή όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα για τους σκοπούς ασφαλείας. Από εκεί πέρα ομω η Μπαρνιέ θα διαπραγματευτεί την κατάσταση για το τι θα γίνει δηλαδή μετά την 31η Δεκεμβρίου του 20. Ε, τελειώνω, τελειώνω. Να πω λοιπόν μόνο ότι για όλους τους ε, α, βλέπω δύσκολο να μην συμφωνήσω με αυτό το οποίο μας ζητά η Κομισιόν. Λόγω της ίδιας της ευθύνης που έχουμε εμείς για την ασφάλεια των πολιτών μας, ακόμη και όταν πρόκειται για το διασυνοριακό έγκλημα και την τρομοκρατία. Λοιπόν, προκειμένου πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μιλούμε για το διασυνοριακό έγκλημα και την τρομοκρατία, επαναλαμβάνω, Μην ξεχνάτε ότι το να μην παίρνουμε τα προφίλ υπόπτων επιτείνει την ανάγκη επικοινωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πραγματικά για, ποιο λόγο ε, δεν θα θέλαμε να συνεχίσουμε την ανταλλαγή με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και κάτι άλλο από όψος ε, δεδομένων. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του ε, της τη Προύμ, κυρίως το κεφάλαιο 6, το άρθρο 6. Απλώς να μου πει κάποιο εάν ε, έχει εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της Προύμ. Αυτό ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ που με, ε, μου δείχνετε κατανόηση γιατί έχουμε μόνο 6,5, μέχρι τις 6,5 χρόνο οπότε παρακαλώ η κυρία Εντεβέλτ να μιλήσει. Έχω μία ε, πρόταση που θέλω να κάνω να συναντηθούμε εδώ οι σκιώδεις για μια συνάντηση που θα κρατήσει ένα λεπτό για να μην μετακινηθούμε. Πιστεύω πως πρέπει να απαντήσω στα όσα είπε η αξιότιμη συνάδελφος για ε, σεβασμό προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως, σέβομαι και αγαπώ τους Βρετανούς και είμαι πολύ ε, που έφυγαν. Αλλά δεν εμπιστεύομαι αυτή τη στιγμή την ε, Βρετανική κυβέρνηση και δεν δείχνουν αυτοί να σέβονται την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που λένε. Δεν καταλαβαίνω τη σειρά των πραγμάτων. Το Συμβούλιο, κατά τη γνώμη μου, ε, τα κάνει ανάποδα τα πράγματα θα πρέπει πρώτα το Ηνωμένο Βασίλειο να δεχτεί τους όρους μας και μετά να τους δώσουμε πρόσβαση. Διαφορετικά πώς μπορούμε να τους πιέσουμε δηλαδή. Αν υποσχεθήκατε επειδή είσαστε πρόσκοποι ε, και δώσατε όρκο θα σας δώσουμε εμείς πρόσβαση για ποιο λόγο. Είναι μια πολύ σύντομη περίοδος χρονική και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι έτοιμοι να δώσουν πρόσβαση τώρα όταν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ε, συμμορφώνεται με τους όρους, πώς θα με πείσετε εμένα να σας εμπιστευτώ εσάς ότι θα αποσύρετε την ε, ε ανταλλαγή αυτή ε, σε κάποιους μήνες ε, αν δεν συμφορθούν. Γιατί είμαι εδώ αρκετό καιρό και πρέπει να σας πω ότι δεν το έχουν κάνει ποτέ στο Συμβούλιο και, στο, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θυμάμαι καμία τέτοια περίπτωση που να έχουν αποσύρει τέτοιου είδους συμφωνία και δεν πιστεύω ότι θα το κάνετε. Και δεν βλέπω και τι κίνητρο δίνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο να δεχτούν τους όρους της πλήρους αμοιβαιότητας και ε, ιδίων προτύπων ε, προστασίας, αν εμείς έτσι καλώς θα του δώσουμε πρόσβαση. Και αν είναι αυτό το μαγικό παιχνιδάκι που πρέπει όλοι να έχουν, γιατί να μην έχουν οι ίδιοι κίνητρο να δεχτούν την, προ... απόλυτη αμοιβαιότητα και ε, το σεβασμό των κανόνων. Δεν καταλαβαίνω γιατί το επιθυμείτε. Εσείς είστε απόλυτα πεπισμένοι πως είναι αξιόπιστο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Τις τελευταίες εβδομάδες μοιάζουμε να ακούμε πως υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να τους εμπιστευτούμε. Και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ίδιο. Εσείς ήδη το 2015 μας είπατε πως το Ηνωμένο Βασίλειο καταπατούσε με άσχημο τρόπο την ε, διακεκριμένη πρόσβαση που έχει στο ε, σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Και τώρα μας ζητάνε να τους πιστέψουν. Να τους πιστέψουμε και να τους εμπιστευτούμε με τα μάτια κλειστά. Ε, όχι. Και ξέρουμε πως δεν έχουν μοιραστεί μαζί μας ε, πληροφορίες για 75.000 περίπου ε, καταδικασμένους εγκληματίες και όταν το ανακάλυψαν ε, ντράπηκαν τόσο πολύ που το κάλυψαν. Και μου λέτε να τους εμπιστευτούμε. Όχι. Πρώτα θα δεχτούν τους όρους μας και μετά να τους εμπιστευτούμε. Ωραία. Η κυρία Ντελμπό Σκόρφιλντ, είστε εκεί. Σας παρακαλώ. Νομίζω πως και εσείς και η Σοφία τα είπατε όλα. Ε, συνεχίζουμε να επιχειρηματολογούμε σαν να μην είχε γίνει το Brexit. χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις δηλώσεις του Μπόρις Τζόνσον, τις οποίες αναφερθήκατε, μοιάζει να μην στηρίζουμε τα όσα είπαμε ότι θα κάνουμε, δηλαδή ότι θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών ε, και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου και μετά στη σχέση μας στο Ευρωπαϊκό, ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο επισκεφθήκαμε την υπηρεσία μας, την Εουλίσα, η οποία είναι αρμόδια για όλα αυτά τα δεδομένα και όταν τους ρώτησαν υπάρχει τρόπος να προστατευθούν από νέες ε, ε, παραβιάσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μας είπαν όχι, βασίζονται όλα στην εμπιστοσύνη. Μα αποδείχθηκε πως δεν μπορούμε να του εμπιστευτούμε. Όχι μόνο δεν το έκαναν, αλλά μας είπαν και συνέχεια μας δήλωναν πως δεν έχουν κανένα σκοπό να ακολουθήσουν τους δικούς μας κανόνες για την προστασία των δεδομένων και δεν έχουν σκοπό να σεβαστούν τα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λένε τώρα. Δεν θα περιμένουν καν να τελειώσει η μεταβατική περίοδος ο συγητής έχει την πλήρη στήριξή μου και αυτά τα οποία η Σοφή είναι πως ε, ε, αντιστρέφουν την σειρά με την οποία θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Το κάρο πριν το άλογο. Εδώ και αρκετή ώρα μιλάμε για την ασφάλεια. Η ασφάλεια δεν είναι μόνο το να προστατευτούμε από τους εγκληματίες και τα υπόλοιπα, ασφάλεια είναι η ασφάλεια των απλών πολιτών να γίνεται σεβαστή η προστασία των δεδομένων τους και ο ιδιωτικό τους χώρος. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ασφάλειας και βαρέθηκα να μιλάμε τα, μόνο για τα υπόλοιπα. Εγώ εδώ εκπροσωπώ τους πολίτες και συμπαθώ τους Βρετανούς εξίσου με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύουμε το υπόλοιπο της ζωής τους, γιατί η προστασία των δεδομένων είναι τεράστιο θέμα. Ο κύριος Μπουσαντέ, ECR. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Νίκολα Προκατσίνη, ο οποίος είναι συντονιστής και τον οποίο αντι καθίστο εξ ονόματος του ECR τασόμαστε υπέρ της θέσης του Συμβουλίου. αυτή είναι η πάγια θέση μας. Τώρα, μερικά άλλα σχόλια ως προς τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και την οδηγία σε σχέση με την δράση των ε, της, ε, σε σχέση με τη δημόσια τάξη, θεωρώ ότι αυτά είναι ε, προμαχώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως, τόσο τα κράτη-μέλη όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Αυτό είναι πρόκριμα για την ασφάλεια των πολιτών μας. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα δεδομένα. Και γι' αυτό ακριβώς το Συμβουλίο μας λέει ότι υπάρχει κίνδυνος ότι από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου να μην ε, πληρωθεί αυτός ο όρος αλλά γι' αυτό υπάρχει και η ρήτρα αναθεώρησης για να σταματήσουμε με αυτή την ανταλλαγή δεδομένων εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συνεργαστεί και δεν μας δίνει στοιχεία για υπόπτους γι' αυτό. Ε, νομίζω ότι όταν μιλάμε με τόσο ωραία λόγια για το κράτος δικαίου ε, ε, δεν μπορέσουμε να, να θέσουμε αυτά τα ωραία λόγια σε εφαρμογή, αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, τότε βρισκόμαστε ενώπιον ενός καινού. Φαίνεται σαν να πρόκειται για μια στρατηγική διαπραγμάτευση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν ισχύει. Γι' αυτό θέτουμε σε κίνδυνο την όλη κατάσταση και δεν βελτιώνουμε την ασφάλεια των πολιτών. Γιατί οι Βρετανοί δημοκρατικά αποφάσισαν να αποσυρθούν. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Συμφωνώ ε, με αυτά που προελέχθησαν από το ECR. Δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα. Θα πρέπει να ενταχθεί αυτή η συζήτηση στην κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών με βάση τη χρήση του χώρου του Σέγγεν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ποια μέτρα ασφάλειας έχουν εφαρμοστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών στοιχείων. Τι έχει γίνει η υπεύθυνη, μάλλον η προεδρεύουσα, μας είπε ότι έχει γίνει μια αποτίμηση, αλλά τα στοιχεία αυτά έχουν αποτιμηθεί μόνο από τη Γερμανία σε σχέση με την ανταλλαγή στοιχείων DNA. Δεν θα ήταν σκόπιμο να έχουμε μια, ένα σημείο διασύνδεσης μέχρι το τέλος του έτους. Τα δικά σας στοιχεία δείχνουν ότι πολλές ε, χώρες δεν έχουν ανταλλαγή στοιχείων DNA ή δακτυλοσκοπικών στοιχείων, ούτε καν μεταξύ τους. Πώς μπορούμε λοιπόν ε, να, την, τα, να τηρήσουμε την προθεσμία με το Ηνωμένο Βασίλειο και ποιο είναι το, ποια είναι η συλλογιστική να παρατείνουμε την κατάσταση πέρα από αυτό το έτος. Η Συμφωνία Προυμ αφορά ανταλλαγή στοιχείων με όλα, μεταξύ όλων των κρατών μελών. Τώρα, ε, εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, τότε θα πρέπει να ανασυνταχθεί το σύστημα. Νομίζω ότι δεν είναι ένα θέμα χρηστής διακυβέρνησης. Ποια θα είναι η προσπάθεια για την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο interface. Άρα δέχομαι αυτά που είπατε κι εσείς. Έχουμε υπερβεί το χρόνο και οι σκιώδεις στη συνέχεια θα συνεδριάσουν εδώ, γι' αυτό είναι πιο πρακτικό, αλλά θέλουν δύο μέλη να παρέμβουν και επειδή παρέμειναν στην αίθουσα θα πρέπει να τους ανταμείψουμε. Να τους δώσουμε λίγα λεπτά χιτβέγγι και η κυρία Ζίπελ, αν δεν κάνω λάθος. Ζητβέγγι, ε, ευχαριστώ. Όλα θα πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα της σημαντικότητας. Αυτό που ε, είναι πρωταρχικό είναι η ασφάλεια των πολιτών έναντι της τρομοκρατίας. Δεν μας ενδιαφέρει αν μας αρέσει ο Μπόρις Τζόνσον, ε, οι θέσεις του, η κυβέρνησή του, έτσι κι αλλιώς ομφαλοσκοπεί θα πρέπει να ανταλλάξουμε στοιχεία. Εμείς έχουμε στοιχεία από εκείνους περισσότερα από ότι το αντίστροφο. Έχουμε την ώρα, το χρόνο να διαπραγματευτούμε μέχρι το τέλος του έτους για το κοινό καλό και τη δική μας ασφάλεια. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος αρέσει σε ποιον και τι σχολίασε. Αυτά δεν έχουν συνάφεια με τη συζήτηση. Η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρναν όλα τα στοιχεία και χαίρονταν γι' αυτό, αλλά ήταν επιφυλακτικοί να δώσουν στοιχεία. Άρα δεν υπάρχει μία ισορροπία. Το να είναι κανείς ε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είδαμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ακολουθούσε τις κανόνες, τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι δεν θέλει καν να πληρεί τους όρους και τις προδιαγραφές της Ευρώπης. Εάν δεν το θέλουν αυτό ως προς την ασφάλεια των δεδομένων, τι θα γίνει με τη μεταφορά δεδομένων. Μιλάμε για προστασία των δικών μας πολιτών εάν επιτρέψουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχει πρόσβαση στα στοιχεία μας χωρίς να έχουμε έλεγχο για το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία στη συνέχεια. Με εκπλήσει το γεγονός ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε δικαιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο για να έχει πρόσβαση στα στοιχεία μας μετά το Δεκέμβριο του 2020. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να δεχτώ. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους. Να μείνουν στην αίθουσα ε, εγώ, της και οι Σκιώδες να αλλά μια στιγμή η, ο, το Συμβουλίο και η Κομισιόν θα του ακούσουμε. Κοιτάξτε, ε, δεν θέλω μαθήματα για την ασφάλεια. Η ασφάλεια με ενδιαφέρει. Η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι κάτι το οποίο παίρνω πολύ σοβαρά. Rule to convey